πρέπει να ξεκινήσουμε πιστεύω γιατί δεν θέλω να καταδαπανίσω χρόνο ο οποίος θα ήταν πολύτιμος στους ομιλητές μας. Τα συνθισμένα καταρχήν έγκριση μέσης διάταξης. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ανακοινώσεις τώρα της ε, Προέδρου. Έχω κάποιες ανακοινώσεις. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το πιο σύντομη. Πρώτα απ' όλα, αύριο το πρωί έχουμε ανταλλαγή απόψεων που προβλέπεται με την κυρία ένα Σαλγάδο, η οποία είναι η πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ, δυστυχώς, δυστυχώς έπρεπε να αναβάλει την παρουσία της ενώπιόν μας και θα σας δώσουμε τη νέα ημερομηνία το ταχύτερο δυνατόν. Σας πενθυμίζω ότι την προσκαλέσαμε βάσει του άρθρου 121,5 των συνδικών και επομένως θα έπρεπε να έρθει να μας εξηγήσει ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με τις συστάσεις για την πολυμερή εποπτεία για την Ελλάδα συγκεκριμένη. Τώρα, αντί να ακυρώσουμε αυτό το σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης που αφορά την επαφή της κυρίας Αλγάδο, εγώ πρότεινα να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χρονικό ε, τμήμα της συνεδριασής μας για να συζητήσουμε τα θέματα της Ελλάδος και άλλα θέματα τα οποία μπορεί να θέλατε να συζητήσετε. Απλώς περιμένω να έχω την ε, απάντηση από όλων των συντονιστών εάν πράγματι τους ικανοποιεί μια τέτοια ρύθμιση. 10 Μαΐου τώρα. Έχουμε έκτακτη συνεδρίαση την ε, Δευτέρα το απόγευμα. Θα ψηφίσουμε και την οδηγία AFM και το πακέτο για την ε, εποπτεία, τα πακέτα, τις εκθέσεις στο πακέτο εποπτείας. Τώρα, όπως ξέρετε, είναι κάπως ε, ογκώδη αυτά τα έγγραφα και παρά το γεγονός ότι έχουν διανεμηθεί τα έγγραφα ήδη, επειδή μάλλον έχουν διανεμηθεί, δεν θα σας τα ξαναδιανύμουμε, αλλά θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής μας και θα υπάρχουν και μερικά έντυπα αντίγραφα στη συνεδρίαση, αν θέλετε να τα αναδυφίσετε, αλλά επειδή ούτως ή άλλως αυτό είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε αποψήλωση εκταρίων δασών, δεν θα τα ξανατυπώσουμε. Επίσης κάνουμε μια έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο την 5η 20 Μαΐου από τις 9.30 μέχρι τις 11.30 το πρωί και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι οι συντονιστές έχουν πάρει λεπτομέρειες σε σχέση με δύο νέα μέλη για την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για τα θέματα στατιστικής και μας ζήτησαν να πούμε εάν εγκρίνουμε αυτά τα μέλη ή όχι. Πρέπει ως 7 Μαΐου να υπάρξει κάποια αντίδραση από τη δική μας μεριά. Ζητάμε μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι της 5ης Μαΐου να γνωρίζουμε τι γίνεται. Τα βιογραφικά τους έχουν διανεμηθεί σε όλα τα μέλη, οπότε μπορείτε να αντιδράσετε αν θέλετε. Τέλος έχουμε το σχέδιο ψηφίσματος για τις ευρείες κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής στα οικονομικά θέματα και οικονομικής διακυβέρνησης. Το θέμα αυτό, ετήσι μιας πολιτικής ομάδος, αναβλήθηκε η εξέτασή του, ετήσι μιας πολιτικής ομάδος και υποστήριξη από δύο άλλες, επομένως το θέμα αυτό θα αντιμετωπιστεί μεταγενέστερα. Μπορούμε όμως να επανέλθουμε στο σχέδιο ψηφίσματος μόνο για τις ευρείες κατευθυντήρες γραμμές οικονομικής πολιτικής. Εάν και το Συμβούλιο αποφασίσει να αναβάλει την εξέταση του θέματο αυτού μέχρι αργότερα. Για το θέμα τη Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, ξέρετε ότι υπήρξε ένα έκτακτο ευρωπαϊκό, υπάρχει ένα έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο για τις, ε, ζών, για τις χώρες του ευρώ και τι χώρε που είναι εκτό τη ζώνη του ευρώ στι 7 Μαου. Λοιπόν, συγγνώμη που σα έχω επιβαρύνει με τόσες ε, ανακοινώσει, Θα περάσω τώρα στο σημείο 3. Σόφι, θες να πεις κάτι, παιδε μου. Εν συντομία, μονάχα για τα πρακτικά ίσως. Είναι κρίμα που δεν έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με την Προεδρία του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ αύριο. Είναι καλό να αναβάλουμε ανταλλαγές απόψεων με την Προεδρία και να συζητάμε αντίθετα μεταξύ μας. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα σε μια κατάσταση η οποία αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα και ενδεχομένω μέχρι ότου η κυρία Υπουργό έχει χρόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι ξεπερασμένο αυτό το θέμα από τα πράγματα. Η ελπίδα μου λοιπόν είναι ότι θα προσπαθήσετε να βρείτε μια λύση με την Ισπανική Προεδρία. Μήπω υπάρχει κάποια χρονική στιγμή στην οποία μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψε. Εγώ σα διαβεβαιώ, λέει η κυρία Μπάου, ότι θα κάνω έντονα διαβήματα. Έχω ήδη κάνει έντονα διαβήματα και θα τα ξανακάνω προ την Ισπανική Προεδρία. Αλλά στο τέλο δεν μπορώ εγώ να τραβήξω με το ζόρι την κυρία Σαλγκάδου να τη σύρω από τα μαλλιά, ούτω ή και έρχομαι λοιπόν και πάλι στο σημείο 3. Είναι το θέμα μας η, η δημόσια ακρόαση για την Βασιλεία 2 και την αναθεώρηση της οδηγίας για την κεφαλουχική επάρκεια. Η λεγόμενη CRD4 είναι η οδηγία αυτή όπως είναι γνωστή στην ε, κοινοβουλευτική μας αργό. Και έχουμε εκθέσεις πρωτοβουλίας που άπτονται αυτής της έκθεσης με εισηγητή συγκεκριμένη περίπτωση τον Όθμαρ Κάρας. Θέλω να χαιρετήσω λοιπόν όλους τους ε, ομιλητές μας. Θα λάβει το λόγο πρώτα ο Στέφαν Βόλτερ, μετά η Μπάρμπαρα Φρόν, ο Άντρεας Τραϊχλ και μετά ο Άντριαν Μπλούντελ Βίγναλ. Δέκα λεπτά ο καθένας θα λάβουν το λόγο, όχι πάνω από δέκα λεπτά και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι θέλουν να θέσουν ερωτήματα παρακαλώ να το αναφέρουν. Και δίνω τώρα το λόγο στον πρώτο μας ε, ομιλητή. Έχω, έχουμε διανύμει τα βιογραφικά τους, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ανάγκη να τους κάνω μακροσχελείς παρουσιάσεις. Ο κύριος Βάλτερ είναι ο Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής της Βασιλείας για την Εποπτεία των Τραπεζών και αυτό φυσικά από μόνο του δικαιολογεί την παρουσία του. Εδώ κύριε Βόλτερ έχετε το λόγο. Um, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα ότι βρίσκομαι εδώ πέρα προκειμένου να σας παρουσιάσω τις εργασίες της Επιτροπής Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία. Βασικό στόχο του προγράμματο μεταρρύθμιση Επιτροπή Βασιλεία είναι καταστήσει το τραπεζικό τομέα πιο ανθεκτικό, προκειμένου να οδηγηθεί σε μεγαλύτερη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη τόσο στο εγγύσιο και στο απότερο μέλλον. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα πριν από την κρίση χαρακτηριζόταν καταρχάς από πολύ μεγάλη μόχλευση όσον αφορά τον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Είχαμε επίσης υπορβηλική αύξηση των πιστώσεων, πολύ χαμηλό επίπεδο εγγυήσεων και υποτιμολόγηση της ρευστότητα και του πιστωτικού κινδύνου. Επίσης δεν υπήρχαν αρκετά επαρκή, αποθέματα ρευστότητα. Επίσης δεν, δεν υπήρχε κατάλληλη διακυβέρνηση όσον αφορά την αντιμετώπιση του κινδύνου και υπήρχαν κάποια συστήματα αποζημίωση τα οποία δεν ήταν καλά σχεδιασμένα. Επίση, δεν υπήρχαν τα κατάλληλα αποθέματα, κατάλληλε προστασίε για τι τράπεζε προκειμένου να προστατευθούν από, τον φιλοκυ... από τη φιλοκυκλικότητα της αγοράς. Επίσης υπήρξε πολύ μεγάλο συστημικός κίνδυνος και πολύ μεγάλη έκθεση και άνοιγμα των τραπεζών σε ιδιαίτερα μεγάλες αντίξουες συνθήκε. συνθήκες. Η κατάσταση αυτή της κρίσης ε, επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι υπήρχε πολύ μεγάλη μόχλευση, ότι δεν υπήρχαν τα απαραίτητα αποθέματα ρευστότητα και ότι δεν υπήρχαν τα κατάλληλα κίνητρα για την ανάληψη κινδύνου. Θα έπρεπε κανονικά τα standards, τα πρότυπα προστασίας των τραπεζών, τα πρότυπα για τα ίδια κεφάλαια να ήταν πιο ισχυρά, πιο απαιτητικά, όπως άλλωστε προτείνει η Επιτροπή μα. Προκειμένου να διορθωθούν λοιπόν τα προβλήματα αυτά, η Επιτροπή τη βασίλεια προτείνει να ακολουθηθούν οι ακόλουθοι στόχοι προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που είχαμε στην περίοδο πριν από την κρίση. Όλοι οι ηλικοί κίνδυνοι θα πρέπει να καλύπτονται επαρκώ όσον αφορά την κατάρτιση του απαιτούμενου κεφαλαίου, των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων, ιδίω όσον αφορά πολύπλοκε διπλοποιήσεις, παράγωγα προϊόντα κτλ. Επίση, θα πρέπει να υπάρχει το απαραίτητο κεφάλαιο ψηλή ποιότητα προκειμένου να μπορούν να καλύπτονται οι ζημίες. Επίση, θα πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρότερο ρόλο όσον αφορά το βασικό κεφάλαιο των τραπεζών και μεγαλύτερη διαφάνεια. Επίση, θα πρέπει να περάσουμε σε έναν συντελεστή μόχλευση στον πυλώνα 1 που να μπορεί να προστατεύσει τις τράπεζες που αυτές ανοίγονται προς τον κίνδυνο. Επίσης, θέλουμε να έχουμε επαρκή προληπτική προμήθεια για τις τράπεζες, καθώς επίσης και τα κατάλληλα κεφαλαιακά αποθέματα, προκειμένου οι τράπεζες να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αντίξωε συνθήκες που αυτές προκύπτουν. Επίσης, χρειαζόμαστε καλύτερα πρότυπα για τη μέτρηση και τον έλεγχο του κινδύνου ρευστότητας. Επίσης, χρειαζόμαστε καλύτερη ρύθμιση και εποπτεία των συστημικά σημαντικών οργανισμών και χρηματοπιστωτικών οργανώσεων. Επίσης, Πρέπει να βασιστούμε καλύτερα στο νέο εποπτικό έλεγχο που προβλέπεται στον πυλώνα 2. Επίση, καλύτερη πειθαρχία τη αγορά χρειαζόμαστε στα πλαίσια του πυλώνα 3, με μεγαλύτερη δημοσιοποίηση του προφίλ ρίσκου των τραπεζών. Επίση, θέλουμε κάποιε προσεγγίσεις πρακτική φύση, προκειμένου να βελτιωθεί η ε, διαχείριση και η εξυγίανση των διατραπεζικών συναλλαγών. Επίσης χρειαζόμαστε κάποια μικρο και μακροπροληπτικά στοιχεία προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε καλύτερα μοντέλα για τις τράπεζες και προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτές. Ένα μεγάλο τμήμα των μεταρρυθμίσεων έχει να κάνει για τι εταιρείε εκείνες και τις δραστηριότητες εκείνες που είναι συστημικές στη φύση τους. Πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι στις κεφαλαικές απαιτήσει, ε, οι οποίες χρησιμοποιούνται στα χαρτοφυλάκια συναλλαγών, Αναφέρομαι σε πολύπλοκες τιτλοποιήσεις, καθώς επίσης και σε υψηλότερα πρότυπα κεφαλαίων τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις συστημικά συσταμικές τράπεζες. Από τη στιγμή που έχει βελτιωθεί το πλαίσιο αυτό και χρησιμοποιείται καλύτερα επιχειρησιακά μοντέλα και καλύτερη αντιμετώπιση του κινδύνου, όλες οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν κεφάλαια υψηλότερου επίπεδου προκειμένου να σε θέση να απορροφήσουν τις ε, ζημίες. Η Επιτροπή επίσης έδωσε ιδιαίτερη σημασία στις συγκεκριμένες συνθήκες εκείνες που υπάρχουν για συγκεκριμένες κατηγορίες τραπεζών όπως οι συνεταιριστικές τράπεζες ε, ή οι τράπεζες καταθέσεων. Είναι σημαντικό όλες οι τράπεζες να έχουν ε, τα απαραίτητα αποθέματα προκειμένου να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν πιο δύσκολε καταστάσει. Θα πρέπει να έχουν τα αποθέματα αυτά τα οποία θα, βοηθήσουν, θα βοηθήσουν τράπεζε να λειτουργήσουν αντικυκλικά και θα αποφευχθεί κατά αυτόν τον τρόπο να γίνει μια διάχυση τη κρίση ή τη αντίξωση κατάσταση στην πραγματική οικονομία. Οι Τράπεζε τώρα έχουν επιστρέψει στο επίπεδο κερδοφορίας που είχαν πριν από την κρίση. Αυτό οφείλεται στην δημόσια υποστήριξη η οποία δόθηκε από τα κράτη κατά τη διάρκεια τη κρίση. Έχοντα λοιπόν αυτό κατά νου νομίζω ότι θα πρέπει να αναμένουμε ότι τα κέρδη αυτά θα χρησιμοποιηθούν τώρα προκειμένου να δημιουργηθούν αποθέματα κεφαλαίου και ρευστότητα και δεν θα πρέπει να δοθούν τα χρήματα αυτά σε μερίσματα, σε μόχλευση, σε μπόνους. Η Επιτροπή τη ε, Βασιλείας ακολουθεί τι προτάσει και τι συστάσει που έκανε το G20 προκειμένου να δημιουργηθούν τα νέα πρότυπα ανθεκτικότητα που θα πρέπει να έχουν οι τράπεζε. Κατά αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί και η γενικότερη εμπιστοσύνη στο σύστημα. Οι υφιστάμενε ελάχιστε κεφαλαϊκέ απαιτήσει είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλέ και δεν μα προστατεύουν από μία νέα κρίση καθότι Πάρα πολλέ τράπεζε εξακολουθούν να έχουν χαμηλά επίπεδα κεφαλαίων και ένα ιδιαίτερο υψηλό ποσοστό μόχλευσης. Για παράδειγμα, ο στελεστή στάθμη αυτή τη στιγμή που υπάρχει για τη μόχλευση είναι τη τάξη του 50 προ 1. Επίση, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο αυστηρό ορισμό όσον αφορά το τραπεζικό κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή πρότεινε να υπάρχουν ε, συγκεκριμένα εναρμονισμένα πρότυπα ρευστότητα, προκειμένου οι τράπεζε να μπορούν για έναν τουλάχιστον μήνα να αντισταθούν σε ε, έντονες πιέσεις και σε αντίξωες συνθήκες. Πρόεδρος, μπορείτε να μιλάτε παρακαλώ πολύ λίγο πιο σιγά. Διαβάστε το κείμενό σας και αυτό ε, καταστά το έργο των πολύ δύσκολο. Η Επιτροπή λοιπόν δημιούργησε μια συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να επιβλέπεται η μεταρρύθμιση την οποία επιθυμεί. Θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των τραπεζών και μεγαλύτερη βιώσιμη ανάπτυξη των τραπεζών. Στις δικασίε λοιπόν αυτέ έχουμε τα ακόλουθα στάδια. Πρώτον, δημόσια διαβούλευση. Οι μεταρρυθμίσεις για το κεφάλαιο και τη ρευστότητα του Δεκεμβρίου έχουν ε, περάσει σε μια διαδικασία αυστηρή δημόσια διαβούλευση, Η Επιτροπή προσπαθεί αυτή τη στιγμή να θεωρήσει όλες τις επιπτώσεις να αξιολογήσει όλε τι επιπτώσει που θα έχουν οι μεταρρυθμίσει τη. Δεύτερον, αξιολόγηση αντικτύπου. Η Επιτροπή κάνει αυτή τη στιγμή μια πλήρη μελέτη προκειμένου να αξιολογήσει τις επιπτώσεις του πακέτου αυτού μεταρρυθμίσεων στον τραπεζικό κλάδο και σε μονοσμένε τράπεζε. Επίσης, προσπαθούμε να κάνουμε μία βαθμονόμηση για τις απαιτήσει σε κεφάλαια και σε ρευστότητα προκειμένου να έχουμε ένα τραπεζικό κλάδο που θα είναι πιο ανθεκτικό. Τέλος, μακροοικονομική ε, μελέτη αντικτύπου κατά τη διάρκεια τη μεταβατική, κατά την περίοδο τη μεταβατική, η Επιτροπή της Βασιλείας καθώς επίσης και η FSB με, σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με την ε, Διεθνή Τράπεζα ε, Διακανονισμών προσπαθούν αυτή τη στιγμή να αξιολογήσουν ε, την επίπτωση που θα έχει το χρονοδιάγραμμα μεταρρυθμίσεων προκειμένου να μην επηρεαστεί η περίοδος ανάκαμψης από την οικονομική κρίση. Θέλουμε να καταφέρουμε να πετύχουμε ένα τραπεζικό κλάδο ο οποίος θα είναι πιο ανθεκτικός στις κρίσεις και θα παρουσιάζει μια βιώσιμη ανάπτυξη θα χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα χρονοδιάγραμμα και μεταβατικέ περιόδου προκειμένου να καταφέρουν οι τράπεζε να εναρμονωστούν με τα νέα πρότυπα χωρί να ε, κάνουμε το έργο του πιο δύσκολο. Προσπαθούμε να καλύψουμε πολλές τράπεζες στον κόσμο, καθώς επίσης και πάρα πολλά τραπεζικά προϊόντα και πολλά επιχειρησιακά μοντέλα. Δεν μπορούμε να πούμε ποιος, ποια θα είναι η αιτία μιας επόμενης κρίσης. Αυτό μπορούμε να κάνουμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να μην οδηγηθούμε στην κρίση αυτή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όλες οι τράπεζες και όλες οι χώρες να ενδυναμώσουν την δεκτικότητα τραπεζικού κλάδου, ιδίως ε, δεδομένης της παγκόσμιας φύσης των ε, τραπεζικών χρηματοπιστωτικών αγορών και την ταχύτητα με την οποία οι συναλλαγές γίνονται και οι αλλαγές συμβαίνουν από τη μια χώρα στην άλλη. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι οι μεγαλύτερες περίοδοι ύφεσης τελικά συμβαίνουν, προκύπτουν όταν ο τραπεζικός κλάδος δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει διαμεσολαβητικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι σχέδεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Um, we'll, all... Σας ευχαριστώ πολύ. Οι ερωτήσεις μετά. Ας περάσουμε στην παρουσίαση της κυρίας Μπάρμπαρα Φρόν από το Σανταντέρ. Ειδική υπευθύνη για την Βασιλεία 2, διαχείριση κινδύνου, ανάλυση κινδύνου και Αυτό θα γίνει παρουσίαση με διαφάνειες. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας πω μερικές από τις απόψεις μας από την ομάδα Σαντέρ για τις συγκεκριμένες αυτές προτάσεις. Θα κάνω και γενικά σχόλια και μετά θα μπω πιο συγκεκριμένα στο θέμα της ε, ε, δυναμικής ε, προστασίας. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες σε όλα τα slides, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αργότερα με την ησυχία σας. Συμφωνούμε με τους στόχους της Επιτροπής Βασιλείας και της Κομισιόν και με την κατεύθυνση που έχει χαραχθεί στα διάφορα τμήματα των προτάσεων. Επίσης, θέλουμε να σας προσάσουμε μερικά βασικά μηνύματα. Πρώτον, αν και ο νέος προτινόμενος κανονισμός προσπαθεί να εντοπίσει και να επιλύσει προβλήματα που εμφανίστηκαν στην κρίση, όπως η τυπλοποίηση, παράγωγα και δάνεια μεταξύ των τραπεζών, δεν απευθύνεται στις βασικές αιτίες της κρίσης ή τουλάχιστον στους κύριους παράγοντες που οδήγησαν στην κρίση. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να βληθεί υπόψη η έλλειψη ελέγχων και ότι ο κλάδος ε, δεν έχει ισχυρή μορφή διακυβέρνηση και εποπτεία όσον αφορά το δημόσιο τομέα. Οι τράπεζες οι οποίες θα πήγαν καλά στην κρίση φαίνεται ότι και αυτές επλήγησαν εξίσου όσο οι άλλες τράπεζες. Αυτό δεν συμφωνεί με τους βασικούς στόχους, μερικούς τους βασικούς στόχους που έχουν θέσει οι ρυθμιστικές αρχές. Δεύτερο, η πρόταση δεν θα πρέπει να τη δούμε μεμονωμένα. Αντίθετα, επειδή έχουμε πολλές επικαλύψεις και πολλές περίεργες ε, επιπτώσεις προς διάφορες κατευθύνσεις, όλα αυτά θα πρέπει να δούμε ταυτόχρονα πριν ληφθεί τελική απόφαση. Αυτό σημαίνει και η επίπτωση στην πραγματική οικονομία, στους καταναλωτές, στην λειτουργία, την καλή λειτουργία των χρηματαγορών, και τη αλλαγή ενδεχομένω του ρόλου που παραδοσιακά παίζουν οι τράπεζες. Ας έρθουμε στο δεύτερο σημείο. Παρακαλώ το επόμενο slide. Θεωρούμε ότι αν περιοριστεί ο κίνδυνος σε μία συγκεκριμένη τράπεζα, η περιοριστική χρήση των προστατευτικών στρωμάτων όσον να τη μπορεί να επηρεάσει τη ρευστότητα και την σταθερότητα της διατραπεζικής αγοράς, ιδιαίτερα σε πιο μικρές χώρες. Έπειτα, οι επενδυτές μπορεί να διστάζουν να επενδύσουν στις τράπεζες σε σχέση με τη μειωμένη απόδοση και το κατά πόσο πληρώνεται ή όχι μέρεσμα. η έμφαση που δίνεται στην υψηλή ποιότητα ρευστότητα και κεφάλαια, αν και είναι κατανοητή όσον αφορά την μέτρα προφύλαξης, μπορεί να δώσει κίνητρα στη συγκέντρωση των κινδύνων και να δημιουργήσει περίεργες ανεπιθύμητες συμπεριφοράς. Αυτό δεν συμφωνεί με τις ιστορικές πρακτικές που θέλουν να μην στηριζόμαστε σε μία ή σε λίγες πηγές όσον αφορά την ε, ρευστότητα. Ο κανόνας να, ε, που λέει να, να είναι οι ίδιοι κανόνες για όλους, αυτό δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Γιατί σχετίζεται με την τοπική νομοθεσία, η φορολογική νομοθεσία κλπ. Όλα αυτά δεν έχουν εναρμονιστεί ακόμα. Στο βαθμό που τις λογιστικές διαφορές υπάρχουν ακόμα, ε, στις κεφαλαιογορές θα υπάρχει διαφορετικό αποτέλεσμα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση έκπτωση από το φόρο σε σχέση με ορισμένα μετοχικά κεφάλαια. Επίσης δεν συμφωνούμε να μπουν οι διατάξεις του grandfathering που θα ε, στρέβλωναν τους ε, ίσους κανόνες για όλους. επειδή οι τράπεζες που παρέχουν στεγαστικά δάνεια δεν έχουν μεγάλη δυνατότητα δράσης και επειδή υπάρχει μια συγκεκριμένη αναλογία μόχλευσης, θα υποχρεώσει ορισμένε τράπεζε να αποχωρήσουν από ορισμένε αγορέ. Το Σανδοντέρ θεωρεί ότι μόνο αν υπάρξει ένα διάλογο γνήσιος μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με έλεγχο των κανόνων, μόνο τότε θα έχουμε τα σωστά κίνητρα και ένα νέο ρυθμιστικό εποπτικό πλαίσιο θα υπάρξει, το οποίο θα καλύπτει τις βλέψεις και των δύο πλευρών, θα αποτρέψει κρίσεις και θα επιτρέπει ταυτόχρονα τις τράπεζες να λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο ίσων κανόνων για όλους. Η αγορά θα διαφοροποιεί μεταξύ των σωστών πρακτικών και των μη σωστών πρακτικών. Μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Και σε αυτό στο κύριο θέμα μου που είναι το σημερινό, το provisioning. Πριν μπω στο τεχνικό μέρος, θα ήθελα να σας εξηγήσω γιατί ένα σύστημα προληπτικό είναι πολύ σημαντικό για τη σταθερότητα της οικονομίας. Η οικονομική δραστηριότητα υπόκειται σε περιοδικούς κύκλους. Έχουμε καλές χρονιές και μπορεί να έχουμε και χειρότερες χρονιές και στροβάρες σοβαρές Γι' αυτό οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν την ε, ε, πρόνοια να αποθηκεύουν το, χειμώνα, για το, το, το, χειμώνα, το καλοκαίρι για να έχουν το χειμώνα. Τι γνωστή ιστορία με το Μυρμή και με το Τζίτζικα. Πρέπει να προετοιμαστούν λοιπόν για τις μέρες των δεινών. Το ισπανικό μοντέλο είναι αυτό που είναι και η εναλλακτική μας πρόταση. Με κάπως διαφορετική μορφή βέβαια. Οι προτάσεις της Ένωσης και του Σανταντέρ. Το επόμενο slide. Αν τα πράγματα είναι τόσο απλά, γιατί έχουμε σύγχυση στη συζήτηση για το θέμα αυτό. Κατ' εμέ υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένας είναι, αν και όλοι οι ενδιαφερόμενοι κατά κάποιο τρόπο θέλουν να υπάρχει αυτή η προληπτική κάλυψη, τα κίνητρα δεν είναι τα ίδια Εξάλλου οι δηλώσει εδώ που είναι στο, στο slide προέρχονται από δηλώσει όλων των διαφορετικών. Αμερικοί θέλουν να λύσουν το θέμα τη κυκλικότητας ε, βάζοντας προμήθειες σε σχέση με δεχόμενε ζημιέ αργότερα. Άλλοι αναγνωρίζουν τις, ε, θέλουν να γνωρίζουν τις ζημιές <coughs> κάπω πιο νωρί λογιστικά. Άλλοι θέλουν να μην έχουμε υπερβολική αύξηση της, ε, του πιστοτικού δυναμικού. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερη αιτία. Η σύγχυση προέρχεται από το ότι το θέμα του συζητάνε είτε άτομα που έχουν εμπειρία βασιλείας δύο αξιολόγηση κίνδυνου και άλλοι που προέρχονται από τον οικονομικό κλάδο. Επόμενο slide. Οι προτάσεις τώρα για το provisioning υπάρχουν πολλές. Θα έλεγα όμως ότι μπορούμε να τις βάλουμε σε τρεις κατηγορίες. Το μία είναι να πάρουμε τους λογιστικούς κανόνες τη εφετερία, τα άλλα προτάσεις με τη βάση την prudential, προληπτική, και το τρίτο μια συμβαστική λύση μεταξύ των δύο προηγούμενων. Αν και είμαστε υπέρ της πρότασης της Κομισιόν, που συμφωνεί και με τους δικούς μας στόχους για ομοιομορφία, απλότητα, διαφάνεια, Ρεαλιστικά πιστεύουμε ότι θα είναι δύσκολο να γίνει αυτό δεκτό αν δεν αλλάξουν τα λογιστικά πρότυπα. Γι' αυτό η τρίτη κατηγορία, κατά τη γνώμη μας, οι προτάσεις Σανταντέρ, θα γεφυρώσουν το χάσμα. Και θα πρέπει να την προσέξουμε αυτή την τρίτη πρόταση. Όπως επίσης και η πρόταση της Βασιλείας, που θέλει να συγχωνεύσει κατά κάποιο τρόπο όλα τα συμφέροντα Κάπω υπερβολικά βέβαια κατά τη γνώμη μας. Επόμενο slide. Η πρεμήθεια αυτή βοηθάει στο να μην έχουμε υπερθέρμανση τη οικονομία και υπερβολική αύξηση των πιστώσεων. Βλέπετε ποιο είναι ο πραγματικός κίνδυνος από ένα δάνειο, από την αρχή του. Και σε ύφεση αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να μην φτάσει η στιγμή που ξαφνικά να, απότομα να πάψουν να δανείζουν οι τράπεζες ή επειδή είχαν μεγάλη ζημιά να μην έχουν κεφάλαια να διαθέσουν. Έτσι ώστε η συμπεριφορά της τράπεζας να μην επιδεινώσει την ύφαση. Και στο επόμενο slide θα δείτε ένα παράδειγμα με νούμερα. Αυτό που δεν θέλουμε να συμβεί, και αυτό είναι το κύριο μήνυμά μας, είναι το διπλό αυτό σύστημα, όπου τα λογιστικά πρωτοπορίζονται από τη μια μεριά, από του μεν και από την Κομισιόν από την άλλη πλευρά. Το παράδειγμα εδώ βλέπουμε τι ανεπιθύμητα αποτελέσματα μπορεί να έχει μια τέτοια δυτή μέθοδος. Τρία σχόλια στο slide αυτό. Πρώτον, δεχόμαστε το να υπάρχουν λογιστικά πρότυπα να δίνουν αληθή και διαφανή στοιχεία για εικόνα της τράπεζας για τους επενδυτές. Σε Σανεντέρ δεν υπήρξε τέτοιο πρόβλημα για τους επενδυτές. Παρότι έχουμε το σύστημα δυναμικής provisioning, το αντίθετο δεύτερον θεωρούμε ότι όσοι έχουν τα πράγματα, η εικόνα δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με τα σημερινά στοιχεία που έχουμε. Και τρίτον, επειδή η πληρωμή του μερίσματος γίνεται αφού ισχύσει provision και από τους δύο ρυθμιστές, μέσω ισολογισμών προς όφελος του εισηγητή, του επενδυτή, είναι η λύση της βασιλείας. Και το επόμενο slide μας δείχνει ότι η καλύτερη λύση, πρόταση, είναι η σύνθετη λύση συγχώνευσης και μεταξύ ρυθμιστικών οργάνων διεθνώς και καλούμε την Επιτροπή της Βασιλείας και την να πάρει τις αποφάσεις για το provisioning αυτό λαμβάνοντας υπόψη και τις άλλες προτάσεις σχετικά με τα buffers. Η απάντηση του κατά πόσον αυτό επηρεάζει τον κύκλο είναι μη ικανοποιητική. Γιατί όπως σας είπα και πριν, ο υπολογισμός ζημιάς λόγω ενός δανείου Έπειτα δεν μπορούν να γίνουν δεχτές προμήθειες πέραν χαρτοφυλακίων Δεχόμαστε μεν λοιπόν τη λύση της σύγκλησης, οπότε η Κομισιόν από τη μια μεριά και αυτοί που εφορήσουν τις λογιστικές προδιαγραφές θα πρέπει να βρουν ένα συμβασμό χωρίς να αφαιρεθεί η δράση όσον αφορά τον κυκλικό χαρακτήρα, αλλά αυτή η συμβαστική λύση θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένους παραμέτρους για τον υπολογισμό του κεφαλαίου, πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή το τονίζω αυτό δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Και η προσωπική μου γνώμη είναι ότι θα είναι ε, μια ιδέα ότι δεν στέκεται ότι ο χαρακτήρας που επηρεάζει τον κυκλικό χαρακτήρα της οικονομίας ότι ελέγχεται. Πρόεδρος. Δέκα λεπτά δεν ήταν πολλά, αλλά ήταν ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπε. Το κύριο Τράιχελ τώρα, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Erste Group Bank. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Και για μένα είναι μια μεγάλη τιμή που είμαι προσκεκλημένος σας σήμερα ένα μέλος του τραπεζικού κλάδου σίγουρα έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις όπου και να είναι προσκεκλημένο σήμερα. Η κρίση που αντιμετωπίσαμε ήταν μια κρίση η οποία δημιουργήθηκε από τον τραπεζικό τομέα και έχει περάσει τώρα σε μια φάση όπου πρέπει να εμπλακούν οι πολιτικοί για να επανεξετάσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο και ε, το πλέγμα που έχουν δημιουργήσει οι ρυθμιστικές αρχές ώστε να εξασφαλίσουμε ότι και στο μέλλον δεν θα επανέλθει μια τέτοια κρίση. Πιστεύω ότι οι πολιτικοί φορείς όπως η G20 έχουν δώσει τρία κύρια καθήκοντα στους ρυθμιστές. Πρώτα απ' όλα, να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στον τραπεζικό τομέα εν γέννη, ώστε τέτοιου είδους κρίσεις δεν θα είναι δυνατές, δεν θα είναι δυνατόν να συμβούν στο μέλλον. Δεύτερον, θα πρέπει να αποκατασταθεί ένα σύστημα αμοιβών και κινήτρων στις τράπεζες ώστε τα στελέχη των τραπεζών δεν θα έχουν κίνητρα να αναλαμβάνουν υπέρμετρους κινδύνους όπως το παρελθόν. Τρίτον, θα πρέπει οι τράπεζες να επανέλθουν στον αρχικό σκοπό ύπαρξής τους, δηλαδή την αποδοχή καταθέσεων από τους καταθέτες και τροποποίηση και μετατροπή αυτών των καταθέσεων σε δάνεια προς την πραγματική οικονομία. Αυτό είναι το τρίτο σημείο αυτό όπου οι ρυθμιστικές αρχές φαίνεται ότι θα αποτύχουν στο εγχείρημά τους. Και εγώ ανησυχώ πάρα πολύ ότι οι πολιτικοί δεν γνωρίζουν τους ενδεχόμενους κινδύνους οι οποίοι μπορεί να προκύψουν για την πραγματική οικονομία εάν η Βασιλεία 3 εφαρμοστεί με τον τρόπο που προβλέπετε τώρα να εφαρμοστεί. Εγώ εκπροσωπώ μια περιοχή που δεν έχει μια ιδιαίτερα ισχυρή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ενεργοί στην Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία και στην Αυστρία φυσικά. Είμαστε τράπεζα λιανικής, δηλαδή λειτουργούμε σε μια περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου δεν υπάρχουν ουσιαστικά χρηματαγορές. Εξασφαλ. Η περιοχή μας βασίζεται μονάχα σε φορείς σαν τους δικούς μας τραπεζικούς φορείς που δέχονται καταθέσεις από 18 περίπου εκατομμύρια πελάτες που έχουμε και τις μεταμορφώνουν σε δανειοδότηση προς τις εταιρείε σε μια περιοχή η οποία δεν έχει και δεν θέλει να έχει χρηματοδότηση από τις κεφαλαίες αγορές. Αν δείτε τους κανονισμούς που προβλέπονται για τη Βασιλεία 3 σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο, κεφαλογικές απαιτήσει, ρευστότητα ή άλλα τμήματα που αφορούν το τραπεζικό τομέα, αυτό το οποίο δεν είναι σαφές, αυτό το οποίο δεν έχουμε κατανοήσει, είναι η ισχυρή διαφοροποίηση μεταξύ τραπεζικών ενεργειών που υποστηρίζουν την πραγματική οικονομία και τραπεζικών ενεργειών που το κάνουν αυτό μόνο έμεσα ή ουσιαστικά ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες. Το τωρινό πλαίσιο δεν έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε τράπεζες όπως η δική μας οι οποίες κατά 80 έως 90% του κόστους τους αποδίδεται στο να δίδονται τραπεζικές υπηρεσίες στο ευρύτερο κενό, η ρευστότητα την οποία προσποριζόμαστε από τους πελάτες μας έχει καλύτερη μεταχείριση από την ρευστότητα που παίρνουμε από τη διατραπεζική αγορά. Πιστεύουμε ότι η δανειοδότηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο μέλλον, μέσω αυτού του ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο δημιουργείται αυτή τη στιγμή, θα είναι πολύ μειονεκτικότερη σε σχέση με την δανειοδότηση εταιριών που έχουν πρόσβαση. Ίσως είμαι υπερβολικός όταν το λέω αυτό, αλλά λόγω της χρονικής πίεσης πρέπει να είμαι λίγο πιο προκλητικός. Η Βασιλεία 3 ουσιαστικά βοηθάει τις τράπεζες επενδύσεων, αλλά όχι τις τράπεζες λιανικής. Και ας μην συζητήσουμε γιατί μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι είναι απόλυτα κεφαλαιόδες. Οι πολιτικοί να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό και να σχηματίσουν μια εμπεριστατωμένη γνώμη για όλα αυτά, ιδιαίτερα η πολιτική η οποία είναι υπεύθυνη για χώρες όπου δεν υπάρχουν εύρωστες κεφαλαίοι αγορές, όπου η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις μικρομεσαίες εταιρείες και θα συνεχίσει να το πράττει αυτό στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να ελεγχθεί αν υπάρχουν πραγματικά κάποια κίνητρα μέσα σε αυτό το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υποστηρίξουν αυτή την ραχοκοκαλιά της οικονομίας στις περισσότερες από τις χώρες στις οποίες εργαζόμαστε, που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε τρόπους με τους οποίους τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα έχουν τα μέσα να υποστηρίξουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το κεφάλαιο το οποίο θα χαθεί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να ανακτήθει με το να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο έλεγχος σε δραστηριότητες συναλλαγών ή σε ενέργειες των τραπεζών στην κεφαλαία αγορά. Μια διαφοροποίηση λοιπόν μεταξύ τραπεζών που εργάζονται πραγματικά προ όφελο τη πραγματική οικονομία και αυτών που το πράττουν μόνο περιστασιακά ή καθόλου αυτή η διάκριση θα πρέπει να είναι πιο ουσιαστική από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή προβλεπόμενο στο σχέδιο για τη Βασιλεία 3. Είναι γεγονό ότι όχι μονάχα οι μικρότερε χώρες στην Ευρώπη, αλλά και χώρες όπως η Γερμανία, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την άμεση δανειοδότηση και η Ευρώπη γενικά έχει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό άμεσης δανειοδότησης έναντι των Πολιτειών. Και είναι αντίστροφη η λόγοι αυτής της δύο υπήρου στις ΗΠΑ. Περίπου 70 με 80% της χρηματοδότησης είναι από τις κεφαλαίες αγορές, ενώ στην Ευρώπη είναι ακριβώς το αντίθετο, 70 με 80% από τις τράπεζες λιανικής. Αυτό το οποίο λοιπόν προβλέπεται στη Βασιλεία 3 δεν είναι μονάχα κάτι που θα οδηγήσει σε μειονέκτημα τις μικρότερες χώρες της Ευρώπης, είναι κάτι που οδηγεί την Ευρώπη γενικά σε μειονεκτική θέση, γιατί η Ευρώπη εξαρτάται πολύ περισσότερο από την άμεση τραπεζική χρηματοδότηση από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πιστεύω ότι είναι πολύ αργά για να αναστρέψουμε αυτή την πορεία, αλλά πιστεύω ότι είναι καιρός τα κοινοβούλια και οι πολιτικοί αυτοί οι οποίοι βρίσκονται κοντά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ασχοληθούν με το θέμα αυτό γιατί το προβλεπόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τράπεζες, μη σκεφτείτε μοναχά τις τράπεζες, οι τράπεζες μπορούν να ζήσουν με οποιοδήποτε λόγο μόχλευσης και κεφαλαίων. Θα κάνουν αυτό το οποίο τους λένε οι ρυθμιστές, αλλά δεν θίγεται τις τράπεζες έμεσα, θίγεται τις εταιρείε που εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση των τραπεζών και την ικανότητά τους να τους παρέχουν δανειοδότηση δεν είναι οι πρόεδροι των τραπεζών που είναι οι σημαντικοί. Είναι οι διευθυντέ των υποκαταστημάτων στην Ευρώπη, οι οποίοι θα πρέπει τα επόμενα δύο-τρία χρόνια να έχουν πράγματι κίνητρα να δανειοδοτούν τι εταιρείε. Τα τελευταία 50.000 ευρώ που δίνετε σε μια εταιρεία, αυτά είναι τα σημαντικά. Αν τα θα τα δώσετε με ένα λογικό επιτόκιο ή όχι. Εκεί λαμβάνονται οι αποφάσει που θα εξασφαλίσουν ότι θα ξαναμπούμε σε μια οικονομική κάρτιση, σε μια οικονομική κρίση. Αυτό είναι ο λόγος λοιπόν για τον οποίο είμαι ενώπιόν σας για να επιχειρηματολογήσω. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρο. Ο τελευταίος μας ομιλητής είναι ο Άντριαν Μπλόντελ Βίγναρ, αναπληρωτής διευθυντής τη της ε, Οικονομικών Θεμάτων και Θεμάτων Επιχειρήν και ειδικό ε, σύμβουλος στον Γενικό Γραμματέα ε, για τι χρηματοοικονομικές αγορέ των ΩΣΑ. Σας ευχαριστώ. Ας περάσουμε στην δεύτερη διαφάνεια, παρακαλώ πολύ. Σας ευχαριστώ καταρχάς που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω στην Επιτροπή σας αυτή. Θα αναφερθώ σε κάποια τεχνικά ζητήματα. Αν δεν καταλαβαίνετε βέβαια πώς λειτουργεί η Βασιλεία, δεν μπορείτε να νομοθετήσετε και για το ζήτημα αυτό. Πρόεδρο, σας παρακαλώ πολύ, υπάρχει διερμηνία, σας ζητάμε να μιλήσετε λίγο πιο αργά. Έχω όμω μόνο 10 λεπτά έχω στη διάθεσή μου, λέει ο μιλητή πρόεδρο. Δεν μπορώ όμω να σα επιτρέψω να μιλάτε τόσο γρήγορα. Το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουμε και βλέπουμε στη διαφάνεια 2 για το σύστημα της Βασιλείας είναι ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία είχαμε ήδη στη Βασιλεία 2. Άρα πρέπει να γνωρίσουμε αν η Βασιλεία 3 λύνει τα προβλήματα αυτά ή όχι. Το σύνολο του μοντέλου της Βασιλείας είναι ένα μοντέλο το οποίο υποτίθεται πρέπει να λειτουργήσει για όλες τις περιπτώσεις και υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα. Καταρχάς, το πρώτο είναι το portfolio invariance, ότι δεν υπάρχει διακύμανση όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο ουσιαστικά θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι ένα δάνειο έχει ένα συγκεκριμένο κίνδυνο, ένα άλλο δάνειο έχει ένα άλλο κίνδυνο. Η επίπτωση όμως στον πρώτο πυλώνα α, δεν λαμβάνεται υπόψη από όλους αυτούς τους πιστοτικούς κινδύνους. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει εντοπιστεί αυτή τη στιγμή στον, στις υφιστάμενες συστάσεις της Βασιλείας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν το 100% του χαρτοφυλακίου σας βρίσκεται στα εργαστικά δάνεια, τότε ε, εμπίπτει στο δεύτερο πυλώνα. Και εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα για το σύστημα της βασιλείας. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά. Επίσης, ε, ένα άλλο στοιχείο είναι ότι ε, υπάρχει ένας ενιαίος αυτή τη στιγμή παράγοντας, που δεν μπορεί να λειτουργήσει όμως για όλες τις περιπτώσεις κινδύνου. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε αυτά κατά νου όσον αφορά τις υποσχέσεις που έχουμε στα πλαίσια του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τι είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ένα σύστημα υποσχέσεων. Εγώ σου υπόσχομαι να σου δώσω αυτό το ποσό και το καθεξής. Έτσι λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι ένα σύστημα υποσχέσεων. Η πιο βασική απέτηση που θα μπορούσε να έχει κανείς είναι οι ρυθμίσεις να μπορούν να ανταποκρίνονται σε όλες αυτές οι υποσχέσεις με τον ίδιο τρόπο οπουδήποτε και να καταγράφονται αυτές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει όμως στην προσέγγιση της Βασιλείας. Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει ένα, μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση εκ των προτέρων όσον αφορά τον κίνδυνο. Δεν μπορούμε δηλαδή εκ των προτέρων να καθορίσουμε το βαθμό του κινδύνου και να εφαρμόσουμε τους συντελεστές στάθμισης. το αν υπάρχει μια νοτροπία πιστώσεων στι τράπεζε ή κυρίω μια κεφαλοχική νοτροπία στι τράπεζε, αυτό ουσιαστικά δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία αν, αν θεωρήσουμε ότι μία εταιρεία λειτουργεί κυρίως με ομόλογα, αν χρησιμοποιήσει το νέο αυτό σύστημα των CDS, των Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνων Αθέτησης, μπορεί να καταφέρει να μειώσει πάρα πολύ τον κίνδυνό της, ιδίως αν αυτός ο κίνδυνος αναλυφθεί από μία άλλη τράπεζα, από ένα άλλο πιστοτικό ίδρυμα. Και αυτό οδηγεί σε αυτό το οποίο ονομάζουμε ρυθμιστικό άρμπιτρα. Ουσιαστικά είναι μια καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτο εποπτείας. Περνάω τώρα σε μια άλλη διαφάνεια της παρουσίασής μου, στην έβδομη διαφάνεια. Στη διαφάνεια αυτή, στα αριστερά, βλέπετε στον οριζόντιο αυτό άξονα τον λόγο που υπάρχει αυτή στη Βασιλεία στον, στην κατηγορία 1 Προσπαθήσαμε εδώ πέρα να δούμε ποιο είναι ο λόγο των ιδίων κεφαλαίων ω προ τα δάνεια για διάφορε τράπεζε σε διάφορε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον κάθε το άξονα βλέπετε τι ζημίε των ε, τραπεζών ε, εκείνων ω ε, ποσοστό των τραπεζικών του περιουσιακών στοιχείων. Θεωρώ ότι η Βασιλεία δίνει εδώ πέρα κάποια στρεβλά κίνητρα. Ουσιαστικά οι τράπεζε με την καλύτερη κεφαλαιοποίηση είναι οι τράπεζε που είχαν τι μεγαλύτερε ζημίε σύμφωνα με τη Βασιλεία. Και εδώ πέρα χρησιμοποιείται απλώς ένας, ένας απλός συντελεστής μόχλευσης προκειμένου να δούμε τελικά τα πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο κεφάλαιο έχει μια τράπεζα, τόσο μικρότερες λογικά είναι οι ζημιές της θα περάσουμε εδώ πέρα στην ένατη διαφάνεια για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικέ αυτέ οι υποσχέσει και ανταπόκριση υποσχέσει. Σύμφωνα με τι προτάσει τη Βασιλεία 3, πιστεύουμε στον ΩΣΑ ότι όντω μπορούν να γίνουν κάποια θετικά πράγματα. Και το πρώτο θετικό το οποίο βλέπουμε είναι η έννοια του συντελεστή μόχλευση. Ο συντελεστή μόχλευση είναι πραγματικά ο πιο σημαντικό παράγοντα στι προτάσει αυτέ. Θεωρούμε ότι το Dynamic Provisioning επίση είναι μια πολύ σημαντική πρόταση. Επίση είναι σημαντικό να υπάρχει ένα απόθεμα κεφαλαίου, δηλαδή σε περίπτωση κρίσης να μπορεί κανείς να έχει περισσότερα κεφάλαια από τα ελάχιστα απαιτούμενα, προκειμένου να καταφέρει να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει σε καμία περίπτωση κανείς να κατεβεί κάτω από το κατόφλι της ελάχιστης κεφαλαϊκής επάρκειας. Και σαφώς θα πρέπει να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τα υποκειμενικά input που γίνονται στο μοντέλο αυτό. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ότι ε, το βασικό πρόβλημα, το βασικό ζήτημα είναι η απώλεια κεφαλαίων στο παρελθόν και ότι δεν είχαν δοθεί τα σωστά κίνητρα μέσω του ρυθμιστικού άρμπιτραζ. Αυτό που είδαμε ουσιαστικά είναι ότι ε, οι τράπεζες χρησιμοποιούσαν παράγωγα προκειμένου να καταφέρουν να μεταμορφώσουν τον κίνδυνό τους και να τον περάσουν σε κάποιον άλλον. Κατά αυτόν τον τρόπο κατάφερναν να αναλάβουν περισσότερο κίνδυνο παρά τις ρυθμίσεις οι οποίες ίσχυαν. Στη διαφάνεια 12, σας το συγγνώμη για τη διαφάνεια αυτή, λέει ο αν δείτε τη διαφάνεια αυτή θα δείτε στο πάνω μέρος ότι οι ελάχιστε κεφαλαϊκές απαιτήσει σύμφωνα με το σύστημα της Βασιλείας Έχετε εδώ πέρα τον κίνδυνο αγοράς, τον λειτουργικό κίνδυνο και τον σταθμισμένο κίνδυνο στο δεύτερο τμήμα της ε, εξίσωσης. Το 8% είναι οι ελάχιστες κεφαλαϊκές απαιτήσει. Αν δείτε τώρα την δεύτερη εξίσωση, έχετε εδώ πέρα τις ελάχιστες κεφαλαϊκές απαιτήσει σύμφωνα με το συντελεστή μόκλευσης. Ουσιαστικά έχει εδώ πέρα έχει το σύνολο των μη σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας. Αυτά τα πράγματα δεν απαραίτητα ισούνται όμως. Αυτό το οποίο συμβαίνει ουσιαστικά είναι ότι ο συντελεστής μόκλευσης θα γίνει μια σημαντική δέσμευση για τις τράπεζες. Οι τράπεζες σε κάθε περίπτωση θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον στελεστή αυτομόχλευσης και να χρησιμοποιούν τελικά παράγωγα, ακόμα και δεν έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια. Μέσω του ρυθμιστικού άρμπιτρας μπορεί μια τράπεζα να καταφέρει να παρακάμψει τις βασικές απαιτήσεις που υπάρχουν για το κεφάλαιο ο συντελεστή ε, μόχλευση τελικά καταλήγει να είναι στο πλαίσιο τη Βασιλεία η ε, ίστατη λύση για τι τράπεζε και θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Και βλέπετε ότι στην τρίτη εξίσωση η, ε, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Μάλλον στην τελευταία εξίσωση βλέπετε να χρησιμοποιείται το ύψιστο ποσοστό κεφαλαίων. Καταλήγουμε πολλές φορές στα ίδια προβλήματα βάσει του συστήματος της Βασιλείας πάντα. Επαναλαμβάνω ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανταποκρινόμαστε στι υποσχέσει που δίνονται στην χρηματοπιστωτική αγορά με τον ίδιο τρόπο. Δεν πρέπει κανεί να μεταφέρει ουσιαστικά τι υποσχέσει από το ένα χρηματοπιστωτικό μέσο στο άλλο. Όσον αφορά τώρα τι προτάσει που γίνονται για τη ρευστότητα. Σαφώ υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία στι προτάσει που γίνονται σχετικά με τα κεφάλαια από τη Βασιλεία. Όσον αφορά όμω τη ρευστότητα και τι σχετικέ με αυτήν προτάσει, θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι να δούμε ποια είναι η σχέση αιτίου-αιτιατού. Ουσιαστικά Είχαμε καταρχά μία κρίση φεργιότητα ή μία κρίση ρευστότητα. Εμεί θεωρούμε ότι είχαμε μία κρίση φεργιότητα. Ουσιαστικά οι πολίτε άρχισαν να ανησυχούν ότι είχαν συναλλαγέ με έναν οργανισμό με ουσιαστικά ιδρύματα τα οποία βρίσκονταν πολύ κοντά στην πτώχευση. Δεν θα πρέπει να αντιστρέφουμε τα πράγματα. Στην Αυστραλία Τη δεκαετία του 1950 και 60 χρησιμοποιούσαμε το σύστημα αυτό το οποίο προτείνεται αυτή τη στιγμή μέσω του συντελεστή μόκλευση και θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να επιστρέψουμε στο σύστημα αυτό. Οι φερέγγιε τράπεζε θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν και ένα μεγάλο ποσοστό ρευστότητα. Και ακόμα και αν διανύουν μια πάρα πολύ σημαντική κρίση, είναι αυτή που διανύουμε τώρα, θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν υψηλό ποσοστό ρευστότητα. Θεωρούμε ότι με τι προτάσει που γίνονται αυτή τη στιγμή επιστρέφουμε στα όσα ίσχυαν στη δεκαετία του 50 και του 60 και δεν βοηθάμε ουσιαστικά ούτε την αγορά του τι τράπεζε. Στι ε, επόμενε διαφάνειε. Βλέπετε κάποια πράγματα όσον αφορά την ε, αγορά ομολόγων. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι αν ακολουθηθεί το σύστημα το οποίο περιγράφεται στη διαφάνεια αυτή, αναγκάζουμε ουσιαστικά τι τράπεζε να διατηρούν στα ταμεία του πολύ περισσότερα μόλογα από ό,τι θα έπρεπε. Επίση, η χρηματοδότηση, την οποία χαρακτηρίσατε αρχικά ω σταθερή, μη σταθερή, πρέπει να σα πω ότι κατά τη διάρκεια μια κρίση είναι πάντα μη σταθερή, να σταθεί η χρηματοδότηση. Και αν ουσιαστικά αναγκάσετε τις τράπεζες να έχουν περιουσιακά στοιχεία χαμηλού κινδύνου, τότε ουσιαστικά μπορεί να τις αναγκάσετε να αναλάβουν και πολύ υψηλότερο κίνδυνο. Νομίζω ότι ξεπεράσατε το χρόνο κάτι ένα λεπτό. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό. Το βασικό μου πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ένα σταθερό καλάθι κινδύνου. Αν αρχίσετε να λέτε ότι το ένα αντικείμενο είναι λιγότερο, περισσότερο επικίνδυνο από το άλλο, οι τράπεζε θα αρχίσουν να πέσουν με τα στοιχεία αυτά και να ανταλλάσσουν μεταξύ του. Και Ήδη βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη ζωηρή αγορά ανταλλαγής tax assets ανάμεσα στις τράπεζες. Είναι σημαντικό λοιπόν να αποφύγουμε να ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι τράπεζες τις υποσχέσεις αυτές που έχουν δώσει στην χρηματοπιστωτική αγορά. Uh, μας είπατε πολλά νομίζω, μας έχετε ε, αναφέρει διαρκέτα. πιστεύω. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο για να θέσετε ερώτημα στους εισηγητές, ο Όθμαρ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Βρισκόμαστε εδώ διότι σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι θέλουμε να παίξουμε το ρόλο που μας αρμόζει μέσα στα πλαίσια της ε, Βασιλείας 2. Μας έχουν κάνει σαφές ορισμένα μέλη του πάνελ ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία είναι ανοιχτά και φαίνεται ότι υπήρξαν και λανθασμένες επιλογές στο παρελθόν. Και ένα από αυτά τα προβλήματα ήταν ακριβώς ο ορισμός του κεφαλαίου των τραπεζών, των κεφαλαιογικών απαιτήσεων που κατά την άποψή μου δίνουν μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση στις τράπεζες που βρίσκονται μέσα στις κεφαλαιογορές από τις τράπεζες ε, Λιανικής. Επίσης υπάρχει το θέμα των ε, ε μετόχων και επίση υπάρχει το πρόβλημα του κεφαλαίου το οποίο πρέπει να διατηρήσει σε απόθεμα μια τράπεζα σε, σε κάποια ορισμένη χρονική στιγμή και φυσικά τίθεται και το θέμα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλω λοιπόν εδώ να σταθώ στον εκπρόσωπο της Επιτροπής ε, Βασιλείας, ο οποίος θεωρεί ότι η απάντηση την οποία δίνει η Επιτροπή του είναι σωστή, πώς αντιμετωπίζεται τις ε, ανησυχίες που ανέφεραν οι άλλοι τρεις ε, ομιλητές σε σχέση με τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Έχετε μελετήσει τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν κάνουμε κάποια διαφοροποίηση μεταξύ των τραπεζών που είναι ενεργές στις χρηματαγορές και των άλλων με τους κανόνες αυτούς. Μπορείτε να εξασφαλίσετε επίσης ότι θα υπάρξει η πλήρης διερεύνηση των επιπτώσεων για την πραγματική οικονομία και κυρίως πώς θα απαντούσατε στα ερωτήματα και τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι άλλοι ομιλητές μας σήμερα. Ωραία, λέει η Πρόεδρος. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε χρόνο να απαντήσουμε όλα τα ερωτήματα κάθε φορά. Ελπίζω ότι έχετε ένα χαρτί και μπορείτε να γράφετε. Ε, υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος ομιλητών μελών του Κοινοβουλίου που θέλουν να λάβουν το λόγο και μετά μπορείτε να απαντήσετε ομαδών όλα αυτά. Έχω τους εξής τώρα στον κατάλογό μου. Mr. Lamberts, um, Vicky Ford, Sven Wolf Swinburne uh, and myself, if anybody else wants. Αν κάποιος άλλος θέλει να θέσει ένα ερώτημα, ας το πει στη γραμματεία Ούντο Μπούλμαν έχει το λόγο. Εγώ μπορώ να υποστηρίξω τον εισηγητή για το ερώτημα το οποίο ετέθηκε προηγουμένως. Εμείς ως Επιτροπή που εμπλεκόμεθα στην ε, νομοθεσία, δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με ένα ορισμό κεφαλαίου που δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγώ δεν θέλω τώρα να σταθώ σε λεπτά νομικά σημεία, δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Εγώ ενδιαφέρομαι για να υπάρχει μια σαφήνεια στους κανόνες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν αυτούς που λειτουργούν στην πραγματική οικονομία, ιδίω αυτού οι οποίοι δημιουργούν θέσει απασχόληση. Αυτό είναι το ουσιαστικό για μα. Μα ενδιαφέρει ότι αυτοί οι φορεί, αυτέ οι επιχειρήσει θα έχουν πραγματική δανειοδότηση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που θέλω να πω. Το δεύτερο θέμα είναι το ερώτημα του πώ μπορούμε να έχουμε τι σωστέ επιλογέ αντικυκλικού χαρακτήρα την σωστή φορολόγηση, τη σωστή, μάλλον όχι φορολόγηση, σωστή κατεύθυνση του χρηματοοικονομικού τομέα, ώστε να μπορεί να λειτουργεί αντικυκλικά η ρύθμιση και να μην διωγγώνει τις ε, διακυμάνσεις στην αγορά. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από, τους, από τα μέλη του πάνελ που έχουν και πρακτική εμπειρία στην, ε, στην αντιμετώπιση τέτοιων μέτρων. Φίλιπ. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω ερωτήσεις που έγιναν από τους συναδέλφους. Μία ερώτηση προς τον κύριο Μπλάντελ. Μας λέει ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούν τα παράγωγα για να αποφύγουν κανόνες. Αν σας κατάλαβα καλά για την επάρκεια κεφαλαίων που είπατε. Έχετε μελετήσει καθόλου το θέμα το τι είναι ανεκτό και μη ανεκτό συναφορά τα παράγωγα και μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό, να απαγορευτούν δηλαδή ορισμένες πράξεις ή παράγωγα. Αυτό θα βοηθούσε να λύσουμε το πρόβλημα στο οποίο αναφερθήκατε, Πρόεδρος. Είχαμε ερωτήσεις από τρεις συναδέλφους, ας δούμε τις απαντήσεις. Καταρχήν, τις μακροοικονομικές επιπτώσεις, ορισμός του κεφαλαίου, αντικυκλική δράση, κατά πόσο είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και πώς μπορούμε να αποφύγουμε το πρόβλημα που δημιουργούν τα παράγωγα. Α ακολουθήσουμε την ίδια σειρά που είχαμε και πριν. Δεν χρειάζεται ο καθένα να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Ο κύριο Βάλτερ πρώτο. Μερικέ ερωτήσει έγιναν στα γερμανικά και δεν είμαι σίγουρο ότι θα μπορούσα να απαντήσω στα γερμανικά γιατί η επάρκειά μου στα οικονομικά γερμανικά δεν είναι τεράστια, γι' αυτό θα συνεχίσω στα αγγλικά. Λοιπόν, πραγματική οικονομία. Καταρχήν έχουμε την καταστροφική δράση στην πραγματική οικονομία, μια κρίση σε σχέση με το κεφάλαιο που υπάρχει. Σας έδωσα νούμερα, όλοι ξέρετε την επίπτωση αυτή. Και οι τράπεζες Υπάρχει ένα χρηματοπιστωτικός μη τραπεζικό τομέα, αλλά οι τράπεζε είναι στο κέντρο του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην κρίση αυτή όλα συγκεντρώθηκαν, αποκρισταλώθηκαν στον, στις και οι τράπεζες δεν είχαν τα μαξιλαράκια που χρειαζόντουσαν για να απορροφήσουν αυτού τα χτυπήματα. Θέλουμε να έχουμε μια νέα κατάσταση όπου να έχουμε μια πιο ισχυρό ανθυρό τραπεζικό κλάδο που να μπορεί να δίνει δάνεια σε μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, να μπορεί να δίνει με συνεχή τρόπο ρευστότητα, αντί να έχουμε αυτό το ξεκίνα σταμάτα, ξεκίνα σταμάτα που έχουμε μέχρι τώρα. Και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το καθεστώς. Έτσι ώστε και μακροπρόθεσμα αλλά και στη μεταβατική φάση να μην βλάψουμε την πραγματική οικονομία. Κάνουμε οικονομικές αξιολογήσεις όχι κατά τράπεζα μόνο, κάνουμε και υποθέσεις. Αν αυξηθεί η, κεφαλαία, η ρευστότητα κεφαλαίου τόσο της 100 σε αυτό το χρονικό ορίζοντα, σε πιο μεγάλο χρονικό ορίζοντα, ποια θα είναι η επίπτωση στην πραγματική οικονομία και κάνουμε τις μετρήσεις, τη μεταβατική περίοδο και την χρονική ροή με τρόπο που να μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα κεφάλαια που υπάρχουν ή αν χρειάζεται εκ μέρους ορισμένων ε, οργάνων ε, να υπάρξει μεγαλύτερη συλλογή κεφαλαίων. Η εντύπωση μου είναι ότι δεν υπάρχει, ε, υπάρχουν μέτρα σε βάρος των μικρότερων τραπεζών. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα αυτών των αλλαγών έπληξαν τις τιτλοποιήσεις, τα παράγωγα, τέτοιου είδους δραστηριότητε για τις πιο μικρές τράπεζες. Το μόνο που τους ζητάμε είναι στους καιρούς ευημερίας να δημιουργείτε αυτά τα μαξιλαράκια, τους προφυλακτήρες για να τους χρησιμοποιήσετε στην περίοδο των ισχυρών αγελάδων. Πάντως τα μέτρα, τα συγκεκριμένα μέτρα, υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν μεγαλύτερους οργανισμούς. Η Μπάρμπαρα. Ένα πρώτο μου σχόλιο ξεχνάμε μερικές φορές ότι οι αγορές των CDS, ε, των swaps και οι τιτλοποίησεις έχουν και τις θετικές πλευρές και ο κίνδυνος συγκέντρωσης αντιμετωπίστηκε με τις τιτλοποίησεις αρκετά και με την χρήση παραγόγων, πιστοτικών παραγόγων, credit derivatives. Χρησιμοποιήθηκε θετικά. Αυτό που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η κατάχρηση όπου υπάρχει. Όχι να μαζί με τα χλωρά, να, μαζί με τα ξερά να κάψουμε και τα χλωρά. Λόγω των νέων κανονισμών για τα κεφάλαια και την τίτλοποίηση και επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι κανονισμοί δεν αφαιρούμε τα CDOs, τα CLOs τα θέματα άρμπιτρας διαιτησίας, όπως επίσης και ο δίκτυς μόχλευσης μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις τράπεζες σε σχέση με εμπορικά δάνεια. Για τα αντικυκλικά μέτρα και πώς τα βλέπουμε εμείς από τη μεριά του Σανταντέρ. Εμείς θέλουμε σταθερότητα σε απροσδόκητες ζημιές και σε λογιστικές ζημιές για μη αναμενόμενες ζημιές και η FSA στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Τράπεζα της Ισπανίας έχουμε κυκλικές προσαρμογές στην περίπτωση που υπάρξει κίνδυνος πρόχευσης Είμαστε υπέρ αυτής της μεθόδου και θα θέλαμε και οι εποπτικές αρχές να το δεχτούν και να δώσουν τα αναγκαία κίνητρα. Για αναμενόμενες απώλειες, ζημιές, αυτό θέλουμε να ισχύσει για όλο τον κλάδο, γιατί είδαμε ότι απέδωσαν στην ισπανική οικονομία. Η προσαρμογή για το CVA είναι ένα νέο στοιχείο προκειμένου να μην υποτιμούμε τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν με βάση την fair value, τη σωστή τιμή, αν έχουμε όμως ένα καλό λογιστικό σύστημα και σωστή διαχείριση, να δούμε τι υπάρχει κάτω από ένα παραγωγό Μπορεί στην περίπτωση αυτή ορισμένα από τα μέτρα που προτάθηκαν να μην είναι καν αναγκαία. Κύριε Τράιχλ, θέλετε να πείτε κάτι. Να σταθώ λιγάκι στο θέμα της ε, πραγματικής οικονομίας. Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί από την Βασιλεία 3. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει τη διαφοροποίηση μεταξύ της καλής και της αρνητικής χρήσης των ε, παραγόγων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για αντιστάθμιση κινδύνων είτε για κερδοσκοπία τα παράγωγα και δεν νομίζω ότι μπορούν να τα διαφοροποιήσουν αυτές τις δύο χρήσεις οι ρυθμιστές. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν το πρόβλημα από μια διαφορετική οπτική γωνία και να επανέλθουμε στο βασικό πρόβλημα της τραπεζικής λειτουργίας. Το πρόβλημα λοιπόν για μένα είναι το απλό γεγονός ότι οι τράπεζες μπορούν να πωλήσουν τον κίνδυνο, να το μεταβιβάσουν τον κίνδυνο τον οποίο αναλαμβάνουν. Στο παρελθόν αυτό δεν ήταν εφικτό. Όταν η οικονομική ανάπτυξη ήταν πιο αργή και οι τράπεζες ήταν πιο ασφαλείς, γιατί οι τράπεζες απλώς έπρεπε να κρατήσουν τον κίνδυνο στα λογιστικά τους βιβλία μέχρι να οριμάσουν τα δάνεια αυτά. Όταν κάνετε ένα δάνειο 15 ετών και ξέρετε ότι σε 15 χρόνια θα έχετε, έχετε ακόμα αυτό το δάνειο, κάνετε ό,τι μπορείτε για να ξέρετε ότι είναι καλό το δάνειο, γιατί άμα είναι λανθασμένη δανειοδότηση, ανεπισφαλής, θα χάσετε λεφτά. Τώρα μπορούμε να δημιουργήσουμε τον κίνδυνο με δανειοδότηση και να τον πουλήσουμε την επόμενη μέρα. Και συνήθω τον πουλάτε σε συμμετέχοντες στην αγορά, οι οποίοι είναι λιγότερο ίσως εξελιγμένοι και γνώστες των πραγμάτων από ότι εσείς ο ίδιος. Από ρυθμιστική λοιπόν έποψη, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να παραχθούν κίνητρα για τις επιχειρήσεις τις τράπεζες να έχουν τα δάνεια ακόμα στα βιβλία τους και όχι να τα ξεφορτώνονται μέσα εισαγωγικά. Γιατί μπορεί κανείς να μετατρέπει τα δάνεια αυτά σε παράγωγα και ουσιαστικά δεν φαίνονται πια στα βιβλία. Μέσα από ένα πολύπλοκο παιχνίδι έχετε καταφέρει να πουλήσετε αυτόν τον κίνδυνο σε κάποιον άλλο. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν δεν το αντιμετωπίζουν οι ρυθμιστές. Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μπλαντνέλ Βίγνερ επανέρχομαι στο σημείο αυτό των παραγωγών και της πραγματικής οικονομίας. Για την πραγματική οικονομία νομίζω ότι πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός γιατί οι τράπεζες δεν δανείζουν τώρα, οι, πίστοση, οι πιστώσεις καταραίουν και όλα αυτά έχουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Δεν πρέπει να αναμίξουμε το θέμα της σωστής ρύθμισης μακροχρόνια και το πώς θα αντιμετωπίσουμε την τωρινή κατάσταση. Ο λόγος για τον οποίο οι τράπεζες τώρα δεν κάνουν διανυδότηση είναι ότι οι επιχειρήσεις που έχουν συσσωρεύσει πάρα πολύ χρέος αυτή τη στιγμή μειώνουν τη μόχλευσή τους και γι' αυτό δεν θέλουν να δανειστούν περισσότερο. Και οι τράπεζες δεν ξέρουν, έχουν αβεβαιότητα σε σχέση με τους μελλοντικούς κανόνες για το κεφάλαιο κεφαλαιοικής επάρχειας στο μέλλον. Δεν θέλουν λοιπόν να εκτεθούν περισσότερο. Κανείς δεν ξέρει πόσο εύρωστη είναι και αυτή η ανάκαμψη. Κανείς λοιπόν δεν είναι έτοιμος να προχωρήσει σε δανειοδότηση και ο ιδιωτικό τομέα ακόμα μειώνει την μόχλευσή του. Επομένω δεν πρέπει να αναμίξουμε δύο πράγματα, θα πρέπει να σκεφτόμαστε, όπω είπε και ο κύριο Βόλτερ, θα πρέπει να σκεφτούμε για το πώς θα μπορέσουμε να προβλέψουμε τις σωστές νομοθετικές ρυθμίσεις για το μακροχρόνιο επίπεδο, αλλά συγχρόνως να έχουμε και μια σωστή αντιμετώπιση για την τωρινή κατάσταση, για τα θέματα των παραγωγών. Το ερώτημα είναι αν θα πρέπει να απαγορευτούν τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, παραδείγματο χάρη. Αυτό είναι ενδιαφέρον ερώτημα. Εγώ δεν θέλω να απαγορεύσουμε τα προϊόντα. Πιστεύω όμω ότι υπάρχουν κάποια ερωτήματα για το πώ θα πρέπει να γίνονται οι συναλλαγέ αυτών των παραγωγών και αν θα πρέπει να αναμειγνύονται τέτοιε δραστηριότητε με την κανονική δραστηριότητα των αγορών. Θα πρέπει η επενδυτική τραπεζική δραστηριότητα να συνδέεται με την παραδοσιακή τραπεζική δραστηριότητα γιατί υπάρχει πράγματι κίνδυνος μόλυνσης όπου οι, οι απώλειες στις κεφαλαγορές μέσω των ε, ε, μεγάλων ομίλων μεταφέρονται και στις εμπορικές τράπεζες. Αν η AIG στις ΗΠΑ είχε ε, χρεοκοπήσει, θα είχε καταρρεύσει ένα μεγάλο μέρος του οικονομικού συστήματος στις ΗΠΑ. Ούτε η Goldman Sachs θα είχε επιβιώσει. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι μία κρίση δεν διονγκώνεται μέσω του συστήματος. Ακόμα και η Goldman Sachs, όπως σας είπα, θα είχε καταρρεύσει. Και επομένω το θέμα της απαγόρευσης των παραγόγων δεν θα πρέπει να έχει να κάνει με τα ίδια τα παράγωγα, αλλά περισσότερο με το τι ακριβώς δραστηριότητε αναμειγνύει κανείς με τις εμπορικές δραστηριότητε. Νομίζω λοιπόν ότι τέτοια θέματα όπως η παροχή ε, εγγυήσεων παραγωγής χάρη από τις τράπεζες για την έκδοση ομολόγων, η η, η όλη ιστορία της παροχής κεφαλαίων, τα κεφάλαια τα οποία πρέπει να έχουν οι τράπεζες ως αντιστάθμιση κινδύνου θα πρέπει ακριβώς να είναι για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους. Αν δημιουργούν παράγωγα τα οποία δεν είναι εύκολα διαπραγματεύσιμα όπως είναι τα εξοχρηματιστηριακά παράγωγα, τότε δεν μπορεί κανείς να εξασφαλίσει αυτή την σταθερότητα. Επίσης, αν κάποιος παίζει στην αγορά, χρειάζεται να κρατάει ένα ε, ένα απόθεμα γιατί μπορεί να αλλάξουν πολύ γρήγορα οι συνθήκες αγοράς. Για μένα λοιπόν το ερώτημα είναι ποιε είναι οι δραστηριότητε οι οποίε είναι επικίνδυνε. Όχι να απαγορεύσουμε τι δραστηριότητε, να εξασφαλίσουμε ότι οι επικίνδυνε δραστηριότητε δεν γίνονται στου χώρου όπου υπάρχει και η κανονική τραπεζική δραστηριότητα. Επανέρχομαι στο ερώτημα του αν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα παράγωγα για να μεταφέρει τις υποσχέσεις των τραπεζών κάπου αλλού, να τις μεταφέρει τις υποχρέωσεις των τραπεζών κάπου αλλού. Εδώ θα θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η καλύτερη μορφή της ρύθμισης. Θα πρέπει να έχουμε απλώς τραπεζικούς τραπεζική ρύθμιση ή θα πρέπει να συνεργάζονται με αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα ασφάλειας. Θα πρέπει να είναι ο ίδιος ρυθμιστής στον τραπεζικό τομέα, στον, με αυτόν στον ασφαλιστικό τομέα. Να μην μπορούν λοιπόν οι τράπεζε να μετακυλήσουν τον κίνδυνο κάπου που υπάρχουν διαφορετικοί όροι ρύθμιση. Και για μένα επίση είναι θέμα τη μορφή των ρυθμιστών. Δεν θα, μπορεί κανείς, θα πρέπει κανεί να κάνει αυτό το λεγόμενο ρυθμιστικό αρμπιτράζ και να μεταφέρει τον κίνδυνο κάπου αλλού. Πρέπει οι ρυθμιστέ λοιπόν να μην είναι στεγανοί μεταξύ του, να μην έχουμε ένα τέτοιο σύστημα και να, μπορούν, να μην μπορούν οι τράπεζε να περιορίζουν με αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο. Νομίζω ότι αυτό μου είπατε να σταματήσω. Ευχαριστούμε πολύ. Βίκη Φόρντ, Βοφ Κλίντς. Και ενδεχομένω να έχουμε χρόνο και για άλλες ερωτήσεις. Βίκη. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή, καθώς επίσης και όλους όσοι οργάνωσαν αυτή την πολύ καλή συνάντηση με τους εξαιρετικούς αυτούς ομιλητές. Μια συνάντηση που μας δείχνει ότι δίστανται απόψεις ε, ακόμα, μολονότι όλοι συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε νέους κανόνες, νέες ρυθμίσεις για τις τράπεζες. Πρέπει βέβαια να προσέχουμε πάρα πολύ τις λεπτομέρειες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Esther Bank που μας ε, τόνισε ποιος είναι ο αντίκτυπο στις ε, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στους πελάτες. Και το ερώτημά μου έχει να κάνει με το χρονοδιάγραμμα το οποίο θα ακολουθηθεί τόσο για την εφαρμογή των κανονισμών αυτών και για το πόσο δεσμευτικές θα είναι. Μας είπατε ότι έχουν αυξηθεί οι ρυθμίσεις αυτές της Βασιλείας για την τυπλοποίηση. Δεν έχει συμβεί όμως κάτι τέτοιο γιατί ακόμα δεν έχει εγκριθεί νομοθεσία για τη Βασιλεία 3 και υπάρχουν ακόμα διστάμενες απόψεις μέσα στις χώρες και στις τράπεζες για το πότε θα καταφέρουν να εφαρμόσουν τη νέα αυτή οδηγία εξαιτίας των επιπτώσεων που θα έχει στη γενικότερη οικονομία. Θα θέλαμε λοιπόν να αναγνωρίζουμε και να καταλάβουμε πώς ακριβώς κάνατε την αξιολόγηση αυτή αντικτύπου πώς θα κοινοποιήσετε προς εμάς, προς τους άλλους, τις, τα πορίσματα της μελέτης αντικτύπου που κάνει η Επιτροπή της Βασιλείας και καθώς περνάμε από την τρίτη στην τέταρτη οδηγία για την κεφαλαιακή επάρκεια, είναι σημαντικό να γνωρίσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητές σας. Ξέρω ότι σε ένα ιδανικό κόσμο θα θέλατε να εφαρμόσετε τα πάντα, όμως δεν ζούμε σε ένα τέτοιο κόσμο, επομένως τι θα εφαρμόσετε πρώτο και με ποιο χρονοδιάγραμμα, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ, Σβέν. Στα γερμανικά. Και βλέπω τον κύριο Λάγκεν, ο οποίος χαίρεται ιδιαίτερα γι' αυτό. Έχω ένα ερώτημα για τον κύριο Τράιχελ. Και άλλοι χαίρονται που μιλάω γερμανικά. Πολύ ωραία. Ακόμα και ο κύριος Μπούλμαν αρχίζει να χαίρεται που ακούει την μητρική του γλώσσα. Θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπε προηγουμένως και ο Ούντο. Στην Επιτροπή μας υπάρχει μια μεγάλη ευαισθησία για την πολυμορφία των τραπεζών στην Ευρώπη και μεταξύ διαφορετικών κρατών επίσης τι διαφορές που υπάρχουν. Και τώρα δυσκολεύομαι να μιλήσω γερμανικά. <laughs> υπάρχει μια μεγάλη ευαισθησία μας ως βουλευτών ώστε η ρύθμιση η οποία θα εφαρμοστεί να μην αφορά μονάχα τις προδιαγραφές της Βασιλείας, αλλά και το πώς θα εξασφαλίσουμε ένα σύστημα εγγυήσεων να υπάρχει μια εξασφάλιση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Εγώ, κύριε Τράχελ, άκουσα πολύ με μεγάλη προσοχή αυτά που είπατε, αλλά έχω τώρα να κάνω και μια ερώτηση. Εσείς είσαστε ένας όμιλος αυστριακός τραπεζών ταμιευτηρίου. Γιατί εσείς ζητάτε τόσο πολύ όμως όταν λέτε όλα αυτά που λέτε. Στην Αυστρία το, το κράτος το οποίο σας έχει υποστηρίξει να μην υποστηρίξει την ε, οδηγία για τα επιτόκια. Νομίζω ότι ε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Αλλά θα ήταν χρήσιμο να έχουμε μια καλύτερη τεκμηρίωση. Γιατί εσείς τώρα υποστηρίξατε ότι η Αυστρία δεν πρέπει να δεχτεί την οδηγία για τα επιτόκια και αν είσαστε, αν μια τόσο συμπαθητική και οικογενειακού χαρακτήρα τράπεζα, γιατί έχετε και μια θηγατρική στις νήσους Καϊμάν. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να σκεφτείτε αν με τον τρόπο αυτό υποστηρίζετε την πραγματική οικονομία, όπως είπατε και εσείς που είπατε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Thank you. Wolf. Ευχαριστώ, Λεπρόεδρος. Παρακαλώ. Λέει ο κύριος Κλίντς. Ένα ερώτημα στον ε, Στέφαν Βάλτερ, τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Βασιλείας. Έχουμε δει ήδη ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτάσεις της Βασιλείας εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ για άλλες δεν υπάρχει μια σωστή εφαρμογή. Το πρώτο μου ερώτημα λοιπόν πώς αυτή τη φορά εκτιμάτε την κατάσταση. αν, μπορέσουμε να πείσουμε, αν θα μπορέσουμε να πείσουμε όλου του εμπλεκόμενου ότι θα εφαρμοστούν αυτά τα νέα μέτρα ή αν θα μείνει πάλι πίσω η Ευρώπη. Το δεύτερο είναι το ερώτημα τη Βίκυ Φόρντ. Εμεί έχουμε πραγματικά διαφορετικέ θέσει εκκίνηση σε ό,τι αφορά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τόσο στην Ευρώπη όσο και στι Ηνωμένε Πολιτείε. έχουμε ήδη μέσα στην Ευρώπη μεγάλη διαφορά μεταξύ της Γαλλίας και της Ισπανίας από τη μια πλευρά και της, μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας από την μια μεριά και Γερμανίας και Γαλλίας από την άλλη πλευρά σε ό,τι αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Και μέσα από αυτές τις διαφορές πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ένα κοινό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Πώς θα ήταν δυνατό να κάνουμε κάτι τέτοιο. Γιατί αυτό θα οδηγούσε σε υπερβολική πίεση σε ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θα πρέπει να τροποποιήσουν σε μεγάλο βαθμό τα τις κεφαλοχικές τους απαιτήσει. Εάν γινόταν αυτή η εφαρμογή, ένα ερώτημα τώρα στον κύριο Μπλάντελ Βίγναλ. Δεν ξέρω τώρα πώς το προφέρει κανείς. Αν είσαστε από την Αυστραλία ή από τη Σκανδιναβία, δεν έχω καταλάβει. Βασίλη Μπλούντελ λέτε. Υπήρξατε πρόεδρος μιας επιτροπής που εκπώνησε μια έκθεση στον ΩΣΑ για τις στρατηγικές εξόδου από τη χρηματοοικονομική κρίση. Εμένα θα με ενδιέφερε μετά από αυτά τα οποία είπατε σήμερα και τα οποία φαντάζομαι ότι προέρχονται και από αυτή την έκθεση. Έρχομαι στην πρόταση που αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο για το πώς θα υπήρχε αυτή η οργάνωση διαμεθοριακών δραστηριοτήτων, χρηματοπιστωτικών φορέων, και πώς θα φτιάχνετε τα λεγόμενα firewalls, τα λεγόμενα φράγματα, <clears throat> ώστε να υπάρξει κάποια αντιμετώπιση των κινδύνων. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα μέσω, αυτών των, μέσω αυτών των μέσων να περιοριστεί ο κίνδυνο. Εξακολουθείτε να υποστηρίζετε ακόμα αυτή την πρόταση του ΩΣΑ που είχατε διατυπώσει εσεί ο ίδιο. Και τέλο, <clears throat> εμένα μου φάνηκε ενδιαφέρουσα η υποκειμενική αυτή αντιμετώπιση που αναφέρθηκε και από τον κύριο τράχλεξαν ότι αυτά, όλα αυτά τα οποία προτείνονται τώρα είναι καινοφανή μέσα στα πλαίσια της, ε, της διαδικασίας της Βασιλείας. Το λέω πολύ προσεκτικά ότι πραγματικά εξεπλάγει γιατί νομίζω ότι είναι, είπατε ότι είναι καινούργια αυτά τα στοιχεία στη διαδικασία της Βασιλείας. Πολύ ωραία, ακούσουμε τις απαντήσεις. Ας ακολουθήσουμε την ίδια σειρά που είχαμε και πριν από λίγο. Κάποιες ερωτήσεις όμως ήταν προ συγκεκριμένους ομιλητές. Ας ακούσουμε πρώτον κύριο Walter. Όπως λέμε στα αγγλικά, δύσκολο το κοινό που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Λοιπόν, ας αναφερθούμε σε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή. Όσον αφορά του κανόνες για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Η Επιτροπή Βασιλείας λέει ότι θα πρέπει να ισχύουν οι σχετικοί κανόνες μέχρι το τέλος του έτους. Θα πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι το τέλος του έτους. Έχουμε κάνει μελέτη αντικτύπου. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μία ακόμα μελέτη λίγο πιο συγκεκριμένη, λίγο πιο λεπτομεριακή, η οποία θα δημοσιευθεί πολύ σύντομα σε ένα-δύο μήνε στα μέσα του έτου, εν πάση περιπτώσει. Και ουσιαστικά εδώ πέρα θέλουμε να γνωρίζουμε αν θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω βελτιώσει όσον αφορά τι κατευθυντήρε γραμμέ για την εφαρμογή των κανόνων αυτών. Εμεί εξακολουθούμε όμω να λέμε ότι θα πρέπει εγκαίρω να εφαρμοστούν οι κανόνε αυτοί. Καταλαβαίνω ότι Ορισμένοι αναφέρονται στι ΗΠΑ που ενδεχομένω να καθυστερήσουν την εφαρμογή. Ήρθαμε σε επαφή όμω σε ύψιστο επίπεδο με του αξιωματούχου των Ηνωμένων Πολιτειών και έχουν και αυτοί δεσμευτεί να εφαρμόσουν του κανόνε αυτού το συντομότερο δυνατό και θέλουν και αυτοί να κάνουν του κανονισμούς αυτού, νόμο αστικά για τη χώρα του. Αναφερθήκατε στη Βασιλεία 2 που δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα και θα πρέπει να περιμένουμε ουσιαστικά για τη Βασιλεία 3 Καταρχά, πρέπει να σας πω ότι είναι σημαντικό πρώτο, πρώτα οι ΗΠΑ Πολιτείες να εφαρμόσουν πλήρω τη Βασιλεία 2. Την έχουν εφαρμόσει ως κανονισμό, αλλά στην πράξη δεν έχει αρχίσει να ισχύει για πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τον Απρίλιο έξι ακόμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ συμμορφώθηκαν. Θα φτάσουμε στα 10 μέχρι τα μέσα του έτους και οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν να αρχίσει να ισχύει για όλα τα ιδρύματα μέσω τη διαδικασία του G20. Όσον αφορά τώρα το κεφάλαιο, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν κάνει συγκεκριμένε δοκιμέ και τεστ και έχουν πολύ συγκεκριμένε απαιτήσει όσον αφορά τον ορισμό του κεφαλαίου και όσον αφορά τα κεφαλοχικά αποθέματα, τα buffers. Έχουν λοιπόν πιέσει πάρα πολύ οι Ηνωμένε Πολιτείε για υψη, υψη, υψηλά κεφάλαια, υψηλή ποιότητα. Όσον αφορά τώρα του λόγου στου οποίου αναφερθήκατε και στο ότι υπάρχουν χώρε που ξεκινάνε από διαφορετικά σημεία κίνηση, πρέπει να σα πω ότι όταν μα χτύπησε η κρίση, άρχισαν οι αγορές να βάλουν κατά των κεφαλαίων της κατηγορίας 1 και υπήρχαν πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία βρίσκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Επομένως, η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει να έχουμε ένα πραγματικά χαμηλό κατόφλι, να μην μπορεί κανείς μεμονωμένα να χειρίζεται το συντελεστή μόχλευσης ή και άλλους συντελεστές θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τον ίδιο τρόπο και με το ίδιο χρονοδιάγραμμα. Όσον αφορά τις προτεραιότητες, Σαφώς χρειαζόμαστε έναν ορισμό του κεφαλαίου, έναν ορισμό του ισχυρού κεφαλαίου, ορισμό και αντιμετώπιση όλων των κινδύνων, αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να αναφερθούμε και στο ζήτημα της ρευστότητας και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως σας είπα πολλά ιδρύματα παρουσιάζονται φερέγγια αλλά στην πράξη δεν έχουν ρευστότητα. Καταλαβαίνετε ότι μακροπρόθεσμα μπορεί να έχουν ρευστότητα αλλά θα πρέπει και κατά τη διάρκεια να έχουν ρευστότητα. Ήρθαμε σε επαφή με πολλούς παράγοντες για τα ζητήματα αυτά και προσπαθούμε πραγματικά να προτείνουμε μια πρόταση που θα λύνει τα πραγματικά αίτια της κρίσης. Θέλουμε να μπορούμε να συμπεριλάβουμε πολλά επιχειρησιακά μοντέλα. Θέλουμε να καταφέρουμε να συνδυάσουμε μικρο και μακροπροληπτικά μέτρα. Έχουμε λάβει πολλές παρατηρήσεις, πολλά σχόλια, τα οποία θα μελετήσουμε πολύ προσεκτικά και θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το πακέτο αυτό μέτρων και προτάσεων ως προς την δομή του και ως προς τη βαθμονόμησή του. Πιστεύουμε πάντως ότι έχουμε κάνει κάποιες κέρυες προτάσεις, τις οποίες αν δεν ακολουθήσουμε ο κίνδυνος θα είναι πάρα πολύ ψηλός. Θα κινδυνεύουμε να ξαναμπούμε σε μια κρίση. Επίσης, τα πράγματα πάντα δεν μας βοηθούν, η συγκυρία δεν μας βοηθά αυτή τη στιγμή. Πολλές φορές ε, ε, οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες, κυρίως ο κόσμος ξεχνά τις παρελθούσες κρίσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να τις έχουμε κατά νου και να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε την κατάλληλη ισορροπία στην αγορά. Δεν μπορούμε όμως αυτή να περιμένουμε, δεν έχουμε χρονικό περιθώριο τριών ετών όπως ακούστηκε. Πρέπει εδώ και τώρα να προχωρήσουμε στις προτάσεις αυτές. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Ας είστε παρακαλώ πολύ σύντομοι στις απαντήσεις γιατί έχουμε ακόμα γύρω ερωτήσεων. Μπάρμπαρα, θέλεις το λόγο. Βέβαια, οι ερωτήσει δεν είναι για μένα ε, ειδικά. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω πόσο είναι κρίσιμο να έχουμε ένα ενιαίο χρονοδιάγραμμα εφαρμογή διεθνώ, διότι οι τράπεζε λειτουργούν σε παγκοσμιοποιημένο επίπεδο. Και είδαμε τι έγινε με τη Βασιλεία 2 όταν οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν την εφάρμοσαν. Δεύτερο, όχι μόνο ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο κανόνα μόνο και στη Βασιλεία 2 δεν είναι, υπάρχει μία Βασιλεία 2, υπάρχουν εκατοντάδες Βασιλείες 2 στην αγορά αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν είναι και πολύ καλό όσον αφορά τη διαφάνεια. Και θα οδηγήσει μάλλον σε περισσότερο αρμπιτράζ. Τώρα, η σωστή χρονική στιγμή για να εφαρμοστούν νέοι κανόνες. Δεν πρέπει να βιαστούμε. Όταν θα δούμε τα αποτελέσματα του ΚΕΡΑΣ θα δείτε ότι πρόκειται για έναν ε, μεγάλη αλλαγή στους κανονισμούς, δηλαδή δεν είναι μικρές αλλαγές, μεγάλες αλλαγές. Και τελικά δεν θα την πληρώσουν οι ένοχοι. Τα τοξικά παράγωγα υπάρχουν ακόμα σε βία πολλών τραπεζών, τελικά όλων των τραπεζών. Καμία δεν εξαιρείται. Γι' αυτό καλύτερα θα είναι να περιμένουμε να γίνει η σωστή κίνηση, μία και καλή, αλλά σωστή να μην χρειάζεται να τα προσαρμόσουμε σε δεύτερη φάση αργότερα. Βέβαια, δεν θα βγουν όλοι από την ύφεση ταυτόχρονα και αυτό μετράει. Και συμφωνώ με τον δίκτυ μόχλευσης όπως αναφέρθηκε. Πρόεδρος, ο κύριος Θα απαντήσω στην ερώτηση του βουλευτή που είπε ότι, τη γερμανικά του, ότι θα μιλήσει σε γερμανικά. Θα το απαντήσω λοιπόν και εγώ στα γερμανικά τα δικά μου. Με ρωτήσατε αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια επίθεση κατά των αυστριακών τραπεζών. Εμείς δεν έχουμε καμία θεατρική καταρχήν στα νησιά Καϊμάν. Είναι πολύ καλά τα γερμανικά σας, αλλά οι έρευνες που κάνατε δεν είναι ιδιαίτερα σωστές. Όπως και άλλες τράπεζες, έχουμε κάποια διεύθυνση στη, στα νησιά Καϊμάν. Αυτό το έχει και η Βαβαρία, αυτό το έχει και η Deutsche Bank. Έχουμε επίσης διευθύνσεις στο Delaware και σε άλλα μέρη του κόσμου για λόγους φορολογικούς. Αν σταματήσουν να υπάρχουν αυτές οι φορολογικές ελαφρύνσεις, δεν θα έχουμε καμία διεύθυνση στα μέτρα αυτά. Και αυτό είναι τόσο απλό. Απλώς θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολλοί οργανισμοί παγκόσμιοι, ακόμα και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, όπως η UNESCO, που χρησιμοποιούν το Delaware σαν ένα τρόπο για να μειώνεται το φορολογικό ε, βάρος. Αν θέλετε μπορείτε να καταργήσετε τα νησιά της Μάχης, αφορολογικούς παραδείσους, το Delaware, τα νησιά Καϊμάν. Αυτό είναι θέμα των πολιτικών, δεν είναι θέμα των τραπεζιτών. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η Πρόεδρος. Ο κύριος Μπλάντερ Βίγναλ. Εγώ θα απαντήσω μονάχα το ένα ερώτημα το οποίο απευθυνόταν σε μένα τον ίδιο. Το θέμα για το έγγραφο που γράψαμε στον ΟΣΑ για τις σταδιοικές εξόδου και ορισμένα ερωτήματα για τα παράγωγα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο λέω σήμερα είναι απόλυτα σύμμορφο με αυτό που είπα στο έγγραφο του ΟΟΣΑ. Όταν εξετάσαμε όλες τις αιτίες των προβλημάτων και τα θέματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν, υπήρξαν κάποιες προτάσεις, οι οποίες πράγματι είναι προτάσεις της Βασιλείας Τρία, τις οποίες εμείς τις υποστηρίζουμε. Αλλά τα δύο θέματα που θέλαμε να απαντήσουμε ήταν ότι χρειάζεται ένας λόγος μόχλευσης χωρίς στάθμιση για να εξασφαλίσει επαρκές κεφάλαιο και δεν, δεν θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται χρήση του κεφαλαίου των εμπορικών τραπεζών σε εκείνο, δηλαδή να γίνει ένας διαχωρισμός για το πού μπορούν να γίνονται ορισμένες συναλλαγές και πού όχι. Αν ενδιαφέρεστε λοιπόν υπάρχει και ένα πολύ καλό έγγραφο το οποίο έχει δημοσιευτεί από την Αυστραλιανή Ρυθμιστική Αρχή για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς τις θηγατρικές και τα υποκαταστήματα μιας ε, εταιρείας holding η οποία η ίδια δεν κάνει τίποτα παρά μόνο παίζει αυτό το ρόλο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο γιατί καλύπτει ορισμένε ρυθμιστικέ πτυχέ. Όταν συζητούσαμε τώρα την πρόταση αυτή και πώ θα κάναμε την, ε, το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων, νομίζω για το, ρόλο, για το λόγο μόχλευση φαίνεται να υπάρχει μια γενική συνένεση. Σχεδόν. όταν πρόκειται για το πώς αντιμετωπίζουμε την δομή των υποκαταστημάτων των ε, θηγατρικών μάλλον, εγώ είχα έρθει σε, σε επαφή και με, την, ε, ε με Σανταντέρ και στην πρότασή μας, το έγγραφο αυτό για τη στρατηγική εξόδου, λέγαμε πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη δομή των, υποκαταστη... των θηγατρικών μάλλον μια μεγάλη εταιρεία και αν θα πρέπει οι θηγατρικέ αυτέ εταιρείε να έχουν καλύτερη προστασία από ότι η υπόλοιπη εταιρεία. Είπαμε ότι σίγουρα μπορεί κανεί να μεταφέρει κεφάλαιο από μια εταιρεία στι θηγατρικέ τη. Και αυτό είναι το σημαντικό θέμα, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν θηγατρικές, το ξέρω. Η τράπεζα λοιπόν αυτή η ευρωπαϊκή είναι μια από τι πιο ε, κερδοφόρες από όλε τις ε, τράπεζες στον κόσμο, κατάφερε να περάσει την κρίση χωρίς μεγάλα προβλήματα. Ένας από τους λόγους που το κατάφερε αυτό ήταν γιατί μπόρεσε να χρησιμοποιήσει τη γεωγραφική διαφοροποίηση και τη δομή των θηγατρικών της εταιρεία. Μια τέτοια δομή λοιπόν μπορεί να είναι καλή. Στην περίπτωση των Banco Santander υπήρξε και καλή διακυβέρνηση. Αλλά το να πούμε να έχουμε μια καλή διακυβέρνηση είναι ότι είναι γεγονός ότι μπορεί να έχει κάνει παραδείγματα καλής διακυβέρνηση αλλά θα υπάρχει πάντα και ένα παράδειγμα καλής διακυβέρνηση. Αν λέτε ναι, πάντα θα έχουμε καλούς προέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου, καλό Διοικητικό Συμβούλιο, τότε είναι καλά τα πράγματα. Αλλά όταν δεν έχουμε, θα πρέπει να έχουμε κάποια νομοθεσία που λέει ότι πρέπει να έχουμε μια δομή με, υπο... με τις που να μην οδηγεί σε κίνδυνο στα κεφάλαια των τραπεζών. Αν δεν αντιμετωπίσετε λοιπόν το θέμα της δομής και βλέπετε ότι Μιλάω παθιασμένα για αυτά τα θέματα που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Αν δεν αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, δεν μπορείτε ποτέ να αντιμετωπίσετε τι κρίσει και αποσύετε τι ευθύνε σα. Δεν πρέπει να επιτρέψετε τι εμπορικέ τράπεζε να εμπλέκονται σε θέματα, σε δραστηριότητε που μπορούν να θέσουν ένα αμφιβόλο το κεφαλαίο του. Και ο καλύτερο τρόπο να το αποφύγουμε αυτό, το έδειξε και η Σαντάντερ, είναι η δομή για τι θηγατρικέ εταιρείε σε μεγάλου ομίλου ανομιγενών δραστηριοτήτων. Είναι καινούργια όλα αυτά. Αυτά τα οποία λέμε σήμερα δεν ξέρω αν εξέπληξαν πολλούς. Οι ιδέες που περιέχονται εδώ νομίζω ότι είναι ιδέες οι οποίες ήδη έχουν ε, δημοσιευτεί και στο παρελθόν. Και το πρόβλημα είναι ότι πάντα όταν βλέπει κανείς το έγγραφο της Βασιλείας 3 είναι ότι περιλαμβάνει πάρα πολλές παραθέσεις από τη Βασιλεία 2. Αν βάλουμε ένα λέει ότι αν βάλουμε ένα συντελεστή 1,25 ή 1,5 θα λύσει το πρόβλημα. Όχι, δεν αντιμετωπίζει τα βασικά προβλήματα που είναι ο λόγος μόχλευσης και ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων για να μην τίθεται ένα αμφιβόλο το κεφάλαιο των τραπεζών. Αν δεν τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα θα έχουμε και πάλι μια κρίση στο μέλλον. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στα μέλη μας. Η ΚΕΙ e έχει το λόγο. ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους ε, ομιλητές μας με πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις και σχόλια. Θα ήθελα όμως να επανέλθω σε κάτι που κατέφθη την περασμένη εβδομάδα στην Ειδική Επιτροπή για την Οικονομική Χρηματοπιστωτική Κρίση, όπου το Policy Department μας έκανε μια, παρουσίαση μια έκθεση με συμπέρασμα ότι στηριχτήκαμε υπερβολικά και για του ε, ρυθμιστέ και για τα χρηματοπιστωτικά δρήματα στη Βασιλεία 2 σε μαθηματικά μοντέλα. Χρήσιμα μεν, αλλά ανεπαρκή σε εποχή κρίσης. Ιδιαίτερα μερικά από τα μοντέλα αυτά δεν έπιασαν πολλούς παράγοντες κινδύνου, όπως η νοοτροπία, γέλης, όρεξη για κινδύνους, αν τους πιάζει ταυτόχρονα όλους αυτούς που είναι στην αγορά. Σε συνθήκες κρίσης και έπειτα όλοι αυτοί οι οργανισμοί και οι ρυθμιστές χρησιμοποιούν πάνω κάτω τα ίδια μοντέλα τα μοντέλα ταυτόχρονα δίνουν την ίδια προστασία κατά κάποιο τρόπο είναι σε βάρο τη ρευστότητα τη αγορά. Και ρωτώ, οι ομιλητέ συμφωνούν ότι υπερστηριχτήκαμε υπερβολικά ενώ σε μαθηματικά μοντέλα. Και ναι, τι μπορεί να γίνει ω προ το πρόβλημα αυτό. Σιλβί. Ευχαριστώ. Ακούσαμε πολλά αγγλικά και γερμανικά. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση στα γαλλικά. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων που γίνεται εδώ, ιδιαίτερα για του πολίτε. Η Επιτροπή Βασιλείας βέβαια δεν υπάρχει για τον πολίτη, δεν ακούει για αυτήν, δεν ξέρει πώς λειτουργεί και τη θεωρεί όχι και πολύ υπόλογη. Χαίρομαι λοιπόν που γίνεται αυτή η συζήτηση γιατί όλα αυτά έχουν επιπτώσει σε όλους μας και με ικανοποίηση σημείωσα την παρατήρηση σας που κάνετε για τις συνεταιριστικέ τράπεζες που στι χώρες της Ένωσης είναι πάνω από το μισό της χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις. Δεν ε, έλασαν το θέμα αυτό. Επειδή κύριε Μπλουν Βινιέλ είπατε κάτι, έχω δύο ερωτήσεις. Όχι μόνο να χρηματοδοτήσουμε την πραγματική οικονομία. Ερωτώ κατά τη γνώμη σας ποιο είναι το καλύτερο μέτρο για να χρηματοδοτούνται μακρόπνοα προγράμματα. Πρέπει να φροντίσουμε η οικονομία μας να προσανατολιστεί προς μια πιο πράσινη και οικονομία. Κατά τη γνώμη σας ποιο είναι το πιο πρόσφορο μέτρο για αυτόν τον προσανατολισμό μακροπρόθεσμα. Και δεύτερη ερώτηση, πάλι προ τον κύριο Μπρούντερ, να δεν έχουν τίποτα με το μοντέλο Σανταντέρ. Σεβαστό είναι, αλλά ερωτώ κατά γνώμη σα, είναι το μοντέλο που είναι το πιο συμβατό με την εσωτερική αγορά, διότι στην Ένωση έχουμε ένα σύστημα που θέλουμε, όχι κατά ανάγκη να υπάρχει σε κάθε χώρα μπλοκαρισμένα, στεγανοποιημένα τα εθνικά κεφάλαια. Πώς το βλέπετε λοιπόν αυτό το μοντέλο σε σχέση με την εσωτερική αγορά που υπάρχει κύριος Τρέζιακ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Μία ερώτηση προς τον κύριο Τράιχελ του Erste Group. Μια πρόσφατη έκθεση του ΩΣΑ λέει ότι τα μπόνους των, τραπεζών, των τραπεζιτών έχουν διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με το από πού προέρχεται η τράπεζα. Αν δίνει δάνεια ή αν είναι μια τράπεζα όπου διανέμει ή πουλάει αυτά τα δάνεια. Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό με, μια σύντομη απάντηση. Πρόεδρος, άλλος συνάδελφος. Κανείς, έχω και εγώ να πω κάτι. και τις αξιολογήσεις επίπτωσης της Βασιλείας. Στις απαντήσεις σας σχεδόν αποκλειστικά μιλήσατε για το χρονοδιάγραμμα, για το χρόνο, μικροεπιπτώσεις, μακροεπιπτώσεις, είπατε, αλλά οι συνάδελφοι και εγώ ενδιαφερόμαστε στο κατά πόσον βλέπει τα πράγματα σε ευρύτερο πλαίσιο. Τι κάνουμε με τις κεφαλαιαγορές, τι κάνουμε με τα παράγωγα, πέρα από τις επιπλέον κεφαλαιοχικές απαιτήσει. Ξέρω ότι η εντολή σας είναι τράπεζες μόνο. Τώρα πια όμως αυτό δεν είναι μεμονωμένο πια. Τον υπάρχουν λοιπόν προφυλακτήρες και μπάφρες για να χρησιμοποιηθούν σε δύσκολους καιρούς, σε περιόδους ύφαση, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή ακόμα είμαστε μέσα σε μια τέτοια κατάσταση. Είμαστε ενδεχομένως στην καλύτερη περίπτωση στην στις αρχές μιας ανάκαμψης. Το να δημιουργούνται λοιπόν προφυλακτήρες, τέτοια και μαξιλαράκια, πώς συντεριάζεται αυτό με την πραγματικότητα που σήμερα ζούμε, που φυσικά είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα, μέλος. Τον έχουμε όμως μια κοινή χρονική γραμμή εφαρμογής, πώς λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις διαφορές. Η Κέι είπε ότι στην προηγούμενη πενταετία του Κοινοβουλίου και πολλοί από εμά μας απασχολούν στο θέμα αυτό του σχετισμού correlations και tail risk. Μας ενδιαφέρει να δούμε το tail risk μέσα στα πλαίσια της Βασιλείας 2 και είχαν γίνει πάρα πολλοί σχόλια σχετικά με παράγοντες ε, συσχετισμού, correlation. Χαιρόμαστε που ασχολείστε με το θέμα αυτό. Αλλά πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα το αντιμετωπίσετε σωστά, θα καταγραφεί σωστά σε σχέση με την τελική επίπτωση που θα έχουν και όχι να τα βλέπουμε σε μια κατάσταση πανικού του τι έγινε πρόσφατα μόνο. Τα μέλη του πάνε καλούνται να απαντήσουν. Αρχίζουμε τον κύριο Γόλτερα. Κύριε Χαρά, θέλετε να... Θέλετε να λάβετε λόγο στο τέλος ή τώρα. Ο εισηγητής θέλει να παρέμβει. Νομίζω ότι το έχει δείξει η συζήτηση πόσο σημαντική είναι η λειτουργία της Επιτροπής μας. Αυτό είναι η εντύπωσή μου και θέλω να το κάνω σαφές. Ότι αν δεν μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματική ισορροπία, αν δεν σκεφτούμε για την τραπεζική δομή, δεν σκεφτούμε για την πραγματική ε, οικονομία της Ευρώπης, αν δεν τα σκεφτούμε όλα αυτά τα πράγματα, θα καταλήξουμε σε αποφάσεις και σε ε, προτάσεις οδηγιών που δεν θα αποσπάσουν καμία πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό πρέπει να πράξουμε όλα τα απαραίτητα από κοινού για να συζητηθούν τα ανοιχτά θέματα και να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα που το υποστηρίζουμε. Και εδώ θα ήθελα να θέσω το ερώτημα. Ποια είναι η αποψή σας για τα θέματα που είναι ακόμα ανοιχτά στην Επιτροπή της Βασιλείας. Πότε θα έχουμε τις, ε, τα πορίσματα της Επιτροπής που αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά. Και επίσης θα υπάρξει κάποια μελέτη που αφορά τον επί, τον αντίκτυπο της κρίσης στην πραγματική οικονομία και ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αν έχετε επίσης και κάποιο σχέδιο χρονοδιαγράμματος για το λεγόμενο trading book, για το ε, χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Είπατε ότι το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών θα πρέπει να κλείνει κάθε χρόνο, στο τέλος κάθε χρόνο. Αλλά ακούμε συγχρόνως ότι οι Αμερικάνοι θέλουν να έχει λυθεί το θέμα αυτό το νωρίτερο στο τρίτο ε, τρίμηνο του 2011 και ίσως και το 2012. Επομένως σημαίνει αυτό ότι μόνο το 12, 2012 θα εφαρμοστεί η, η οδηγία για την κεφαλαιοχική επάρκεια 4 και ακόμα και για την 3 δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πώς συνδέονται μεταξύ τους τα χρονοδιαγράμματα εσείς λέτε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν οι προτάσεις αυτές των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της κρίσης. Καλό είναι αυτό, αλλά συγχρόνως εμείς θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο αυτές οι προτάσεις αντιμετωπίζουν επαρκώς την κρίση και ποιες κυρίως θα είναι οι επιπτώσεις που θα έχουν στην πραγματική οικονομία. Και δεν πρόκειται μονάχα για την αύξηση της ε, κεφαλουχικής επάρκειας, αλλά το πώς αυτή η αυξημένη κεφαλουχική επάρκεια θα προκαλέσει αποτελέσματα μέσω της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Δομής και στην οικονομία. Την προηγούμενη εβδομάδα μας είπανε ότι η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να τηρήσει τους ορισμούς για την κεφαλουχική επάρκεια και ουσιαστικά δημιουργήθηκε μια ανισότητα μεταξύ των τραπεζών που λειτουργούν στις κεφαλαιαγορές και αυτών που δεν ασχολούνται με τις Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα της διαφοροποίησης μεταξύ των τραπεζών επί του βάση του αν συμμετέχουν στις κεφαλαιαγορές και δεν μπορείτε να λέτε ότι θέλετε να έχετε μία ε, ισότιμη βάση ανταγωνισμού όταν τα μέτρα σας ουσιαστικά δημιουργούν αυτήν την ε, διαφοροποίηση μεταξύ των τραπεζών διότι δίνουν μια πιο ευνοϊκή ε, μεταχείριση στις τράπεζες που είναι εγγεγραμμένες στα χρηματιστήρια και συμμετέχουν στα χρηματιστήρια. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι συστηματικές διαφορές μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς στην Ευρώπη έχουμε περισσότερο κεφάλαιο μέσα στις τράπεζες. Υπάρχει περισσότερο ξέρω κεφάλαιο στις τράπεζες, το οποίο σημαίνει και μεγαλύτερους κινδύνους. Αλλά είναι τα μέτρα αυτά τα οποία αναφέρεται για την Βασιλεία 3 ε, είναι πολύ πιο δύσκολο να εφαρμοστούν στην Ευρώπη από ό,τι σε άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ που έχουν ένα διαφορετικό σύστημα σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ, και η πρόεδρος. Επαρέχομαι στον κύριο Βόλτερ. Νομίζω μέχρι τις 5 και 10 μπορούμε να πάμε. Γιατί τα άλλα θέματα στην μέρα διάταξη δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τόσο πολύ χρόνο. Κύριε Βάλτερ, λοιπόν, έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω, λέει ο κύριο Βάλτερ. Είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά τα θέματα και πολύ σημαντικά και έχουμε πολύ λίγο χρόνο να τα διεξέλθουμε. για την εξάρτηση από υποδείγματα, από μαθηματικά υποδείγματα. Είναι γεγονός αυτό. Δυστυχώ δεν έχω να σας δώσω μια απλή απάντηση, δεν έχουμε ένα απλό μοντέλο. Έχουμε συσχετισμούς οι οποίοι κάνουν πολύ πιο πολύπλοκα τα μοντέλα. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να έχουμε πολλαπλούς τρόπους για να βλέπουμε το ίδιο πράγμα, πολλαπλού τρόπου να αντιμετωπίζουμε με ε, δοκιμασία αντικσών περιστάσεων, με λόγους μόχλευσης, με στάθμιση κινδύνου. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μονάχα σε ένα μοντέλο πραγματικά για τη ρευστότητα. Αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο. Σε ό,τι αφορά τώρα την προώθηση μιας πιο μακρόπνοης αντιμετώπισης και σχεδίων τα οποία στο μακροπρόθεσμο θα υποστηρίξουν την οικονομία και το περιβάλλον, και σε αυτή πάλι την περίπτωση νομίζω το να έχουμε πιο σταθερές δομές στον τραπεζικό τομέα που να έχουν πιο μακροχρόνιο χαρακτήρα και που να υπάρχουν και τα κατάλληλα κίνητρα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και όχι μοναχά αντιμετώπιση των τρεχόντων συνθηκών και σκασίλα μας για το μέλλον. Νομίζω ότι υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι προτάσεις, η υπερκυκλικότητα, οι αμοιβέ των στελεχών, όλα αυτά τα θέματα, όλες οι προτάσεις αυτές ελπίζω θα μετακυλήσουν την έμφαση προς ένα πιο ε, βιώσιμο και μακροχρόνιο τρόπο τραπεζικής λειτουργίας. Πρέπει να λάβω υπόψη και το ευρύτερο πλαίσιο, τα αποθέματα ασφαλείας και εδώ λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τις απαραίτητες διασυνδέσεις μεταξύ των πληροφοριών και των στοιχείων που έχουμε συλλέξει τον Ιούνιο-Ιούλιο, να υπάρξει αυτή η σύγκληση όλων αυτών των στοιχείων, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σωστά σταθμισμένο σύνολο προτάσεων που να επιτυγχάνει αυτά που θέλουμε να επιτύχουμε και να αντιμετωπίσει τις αντιρρήσεις και τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί εδώ. Το σημαντικό είναι το QIS, να δούμε πώς αυτό θα μπορέσει να αντιμετωπίσει διαφορα... επιχειρηματικά υποδείγματα, διαφορετικές τράπεζες και σε ποιο βαθμό θα αυξήσει το, τις κεφαλογικές ε, απαιτήσει σε σχέση με την τωρινή κατάσταση και πού θέλουμε να καταλήξουμε, ποιος είναι ένας σωστός ε, σωστός προορισμός για όλα αυτά τα θέματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια, να καταλάβουμε ότι έχουμε μια προσέγγιση αρκετά διαφορετική από την προηγούμενη της Βασιλείας 1 παραδείγματος χάρη και να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι πραγματικά σημαντικό και θετικό αναφέρεται το θέμα των διαφορετικών τραπεζών. Υπάρχουν αυτές που είναι συνεργατικού χαρακτήρα, ενώ άλλε δεν είναι. Αν επανέλθετε στη συμφωνία του Σίδνεϊ το, 2000, το 1999 δεν λέει τίποτα για τις συνεργατικές τράπεζες. Λέει ότι έχουμε απλώς το κεφάλαιο και τα ε, διακρατημένα κέρδη. Αυτό είναι η κεφαλογική βάση. Αλλά τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο αρχών. Πώς θα αντιμετωπίσουμε άλλα μοντέλα ε, τραπεζών. Είδαμε ότι ορισμένε από αυτές τις αρχές, τις 14 αρχές, μπορεί να μην εφαρμόζονται σε αυτή την περίπτωση. Και ορισμένες ομάδες όπως το ΣΕΤΣ μπορούν να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά για να δούμε πώς τι σημαίνει αυτό το πράγμα στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί η Επιτροπή της ε, Βασιλείας έχει 27 χώρες, αλλά το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε έναν τρόπο να εξασφαλίσουμε την ισορροπία στα θέματα αυτά. Όταν μιλάμε επίσης για τα είδη κεφαλαίου, νομίζω ότι μιλάτε για τους σιωπηλούς εταίρους. Εδώ νομίζω το κύριο δίδαγμα από την κρίση είναι ότι αν υπάρχει μεγάλη πίεση σε ορισμένου χρηματοπιστωτικούς φορείς, η αγορά κοιτάζει να δει πόσο κεφάλαιο υπάρχει εκεί για να απορροφήσει τα κτυπήματα και βλέπει ακριβώς την, ε, τις υποτιμήσεις σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο και την αξία αγοράς και εκεί πέρα έχει μεγάλη σημασία το να υπάρχουν διακρατημένα κέρδη. Και αυτά λοιπόν παίζουν σημαντικό ρόλο για να εξασφαλίσουμε την ακαιρεότητα του συστήματος. Οι συσχετισμοί και οι κίνδυνοι σπανίων γεγονότων και εκεί πάλι Συμφωνώ μαζί σας και έκανα ορισμένε προτάσεις για το πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Τα αποθέματα ασφαλείας και η μετάβαση στα νέα πρότυπα. Λέμε ότι πάρα πολλοί φορείς αυτή τη στιγμή έχουν σημαντικά αποθέματα ασφαλείας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι κίνδυνοι οι οποίοι προκύπτουν, αλλά θα ήταν κρίμα αν ο τραπεζικός τομέας δεν ξεκινούσε ήδη από τώρα να κινείται προς υψηλότερα αποθέματα ασφαλείας για να είναι προετοιμασμένο για οτιδήποτε μπορεί να προκύψει. Γι' αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικό και για μας να συμπληρώσουμε το πακέτο μας ώστε να έχουμε μια σαφή κατεύθυνση για τον χρηματοπιστωτικό τομέα ώστε να μπορέσει να κινηθεί προς κάποια θετικά αποτελέσματα. Μπάρμπαρα. Καταρχάς, όσον αφορά την εσωτερική αγορά, ως λιανική τράπεζα θεωρούμε ότι ο, τραπεζικό, ο τραπεζικός όμιλος Σαταντέρ μπορεί να συμμορφωθεί πλήρως με τις συστάσεις που γίνονται. Είμαστε ικανοποιημένοι με τις προτάσεις αυτές. Αυτό που λέμε βέβαια είναι ότι συμμορφωνόμαστε χάρη της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης και της εσωτερικής συμμόρφωσης. δεν σημαίνει ότι το, το μοντέλο του για μας θα μπορούσε να λειτουργήσει σωστά και για άλλες επιχειρήσεις και για άλλες τράπεζες. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα αυτό, ότι εξαρτώμαστε πάρα πολύ από μαθηματικά μοντέλα, νομίζω ότι υπερβάλλουμε εδώ πέρα συχνά. Σε πολλές τράπεζες νομίζω ότι τα μοντέλα οικονομικού κεφαλαίου έχουν λειτουργήσει σωστά. Ο κίνδυνος ρευστότητας που οδήγησε, στην, που σε πτώχευση κατά τη διάρκεια της οικονομικής αυτής κρίσης ήταν ένας κίνδυνος που έχουν αναγνωρίσει οι τράπεζες και που και στο παρελθόν και είπαν ακριβώς ότι τα μοντέλα για τα κεφάλαια δεν μπορούσαν να καλύψουν τον κίνδυνο αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι οι τράπεζες ήταν ειλικρινείς και ανοιχτές. Όσον αφορά τα μοντέλα rating, στον όμιλο Σαταντέρ χρησιμοποιούμε διάφορα από τα, διάφορους από τους δείκτες και τους τελεστές που προβλέπονται από την Επιτροπή της α, Βασιλείας και θεωρώ ότι έχουν λειτουργήσει σωστά. Βέβαια, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε μοντέλο έχει και τους περιορισμούς του και κάθε φορά που συζητάμε για τα μοντέλα, είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιούμε τα μοντέλα αυτά. Αν πρέπει να δείξει κανείς πειθαρχία και χρηστή εταιρική διακυβέρνηση, τότε νομίζω ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς σωστά τα μοντέλα χωρίς να υπάρχουν πολλές πιθανότητες ή πολλά περιθώρια αποτυχίας. Και πάλι αυτό έχει να κάνει με τη χρηστή λοιπόν διακυβέρνηση και τη διακυβέρνηση δεν μπορεί κανείς να την εξασφαλίσει μέσω ρυθμίσεων. Νομίζω ότι η χρηστή διακυβέρνηση καθορίζεται, εξασφαλίζεται μόνο μέσω της εποπτείας. Μόνο μέσω εποπτείας μπορούμε να έχουμε τη χρηστή διακυβέρνηση που επιθυμούμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω και εγώ με τα μαθηματικά μοντέλα. Συμφωνώ πλήρω με αυτό που είπαν και οι προλύσαντε, ότι υπερβάλλουμε πολλέ φορέ να συζητάμε για τα μαθηματικά μοντέλα και οι τράπεζε ε, δεν λειτουργούν πολύ συχνά βάσει των μοντέλων αυτών. Αν θέλετε βέβαια να κάνετε τώρα μια κατανομή της ευθύνης, όσοι πήρανε το βραβείο Νόμπελ για την οικονομία ενδεχομένως να κινδυνεύουν να το χάσουν αν καταπιαστούν με το ζήτημα της Βασιλείας 2 και το ζήτημα της Βασιλείας 3. Όσον αφορά τώρα τα μπόνους, νομίζω το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Είμαστε μία τράπεζα λιανικής, έχουμε 5.000 ε, εργαζομένους, εκ των οποίων 4.700 περίπου λαμβάνουν ένα μπόνου στις τάξεις των 3, 4 ή 5.000 ευρώ. Και είναι ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι παρέχουν τα δάνεια. Και ο λόγος για τον οποίο δεν τους δίνουμε τεράστια μπόνους είναι επειδή δεν κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά κάνοντας, τα... κάνοντας την άμεση αυτή δανειοδότηση. Ουσιαστικά είναι οι τραπεζίτες από τις επενδυτικές τράπεζες αυτοί οι οποίοι καταφέρουν να εξασφαλίσουν πολύ μεγάλα μπόνους ακριβώς επειδή τα δάνεια τα οποία παρέχουν είναι πάρα πολύ μεγάλη αξία. Θα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι αυτοί που παρέχουν τα απλά καθημερινά δάνεια δεν κερδίζουν πολύ ψηλά μπόνου και έχουν επηρεαστεί και αυτοί από την κρίση και από τη γενικότερη κοινή γνώμη εναντίον των τραπεζών αυτή τη χρονική περίοδο. Και βέβαια το πρόβλημα αυτό είναι πολύ μεγάλο και πρέπει να επιληθεί. Όσον αφορά τώρα τα αποθέματα ασφαλείας. Δεν θα ήθελα να κάνω μια πολύ μεγάλη διαφήμιση σήμερα για την Ισπανία. Ήδη μίλησε η συναδελφός μου για την Σαταντέρ. Πάντως αυτό έχει να κάνει με το πόσο συστημικά σημαντική είναι μια τράπεζα και εμεί χρησιμοποιούμε το ίδιο μοντέλο με τη Σαταντέρ. Και όταν ήρθα στην ε, αίθουσα αυτή σήμερα για την συνάντηση, υπήρχαν ορισμένοι από τους συναδέλφους εδώ πέρα στο πάνελ που δεν ήξεραν καν, ο κύριος Μπλάντελ για παράδειγμα, ότι εμείς υφιστάμεθα ως τράπεζα. Πάντως παρόλα αυτά ας μιλήσω για το buffering, για τα αποθέματα ασφαλείας, ζήτημα εξίσου σημαντικό. Ο τρόπος με τον οποίο διαρθώ, διαρθρώνεται σήμερα ενδεχομένως να λειτουργήσει καλά κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή όμως, επί του παρόντος, θέτει το επίπεδο κεφαλαίου στο επίπεδο εκείνο που απαιτείται από τα αποθέματα ασφαλείας. Ενδεχομένως ε, το ποσοστό να είναι 6%. Αν θέλετε όμως να δώσετε μέρισμα στους μετόχους σας, θα πρέπει να πάτε στο 9%. Ή διαφορετικά θα χάσετε ουσιαστικά τους μετόχους, οι οποίοι θα γνωρίζουν ότι θα είναι σε θέση να λάβουν μέρισμα αν δεν χρησιμοποιήσετε αυτό το υψηλό ποσοστό. Και το αντίθετο βέβαια ισχύει μέσω των αποθεμάτων αυτών ασφαλείας τα επομενα δυο δύο-τρία χρόνια οι τράπεζες που δεν έχουν μετοχικό κεφάλαιο, οι τράπεζες που, έχουν, που δεν έχουν μετόχους ή που έχουν μετόχους που δεν ενδιαφέρονται για λήψη μερισμάτων βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση. Και βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επικρίνει αυτού του είδους την διοργάνωση των τραπεζών. Υπάρχουν τράπεζες οι οποίες έχουν μετόχους που δεν ζητάνε μερίσματα, επομένως δεν ασχολούνται καθόλου με το ζήτημα του buffering, με τα αποθέματα ασφαλείας. Νομίζω ότι η Ισπανία έχει καταλήξει σε ένα πολύ καλό σύστημα αντικυκλικού provisioning. Για ποιο λόγο να μην κάνουμε και εμείς το ίδιο έχει ευνοήσει ιδιαίτερα το ισπανικό τραπεζικό σύστημα, αποτελεί ένα από τα σημεία του ισπανικού τραπεζικού συστήματος. Σας καλώ λοιπόν να το αντιγράψουμε με τον ένα τον άλλο τρόπο από το να επινοήσουμε κάτι καινούριο. Um, Ευχαριστώ πολύ. Και τέλος, ο τελευταίος ομιλητή μας. για τα μαθηματικά μοντέλα οι υποθέσεις, μάλλον το πω αν γνωρίζετε για τα μαθηματικά μοντέλα που υπάρχουν κάτω από το σύστημα της βασιλείας, πριν να διαβάσετε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο του Federal Reserve πριν από χρόνια που αναλύουν τα μαθηματικά στοιχεία του μοντέλου αυτού. Δηλαδή το όλο σύστημα έχει γίνει για κρίσεις τραπεζών που δημιουργούν από ένα παγκόσμιο κίνδυνο, να έχουμε έναν ιδιάζοντα κίνδυνο σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή προϊόντα σε μια συγκεκριμένη χώρα, η Βασκία δεν έχει να σα πει και πολλά πράγματα. Και αν δείτε του συντελεστέ συσχετισμού, α πούμε, το αυξήσουμε κατά 1,15% διότι στο συσχετισμό διαπιστώθηκε αυτό, κάντε την προσαρμογή. Είναι σαν να δίνετε μάχε παρελθόντο. Τα πράγματα είναι τελείω διαφορετικά. Ο συντελεστέ οι παράμετροι μπορεί να είναι όλα διαφορετικά, συντελεστέ κλπ. Τα μαθηματικά στηρίζονται σε φυσιολογικά μοντέλα και ξέρουμε ότι στις χρηματοπιστωτικές αγορές τα φυσιολογικά δεν ισχύουν. Τι να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Ναι, να υπάρχουν τα μοντέλα αυτά και είμαστε υπέρ των άλλων ε, μεθόδων επίσης, όπως το συντελεστής μόχλευσης που δεν απαιτούν μαθηματικά μοντέλα, συστήματα μετρήσεων και να υπάρχει κάποια ποινή για τη συγκέντρωση κατά των αποκλήσεων από ένα βασικό κριτήριο μέτρησης benchmark που ισχύει. Αυτό θα ήταν μια καλύτερη λύση. Τώρα, για τις γαλλικές ερωτήσεις. Τι πρέπει να κάνουμε για τον μακρόπνο, μακρόπνη χρηματοδότηση είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος διακυβέρνησης διαχείρισης των επιχειρήσεων, corporate governance. Ξέρουμε ότι ο ΣΑ έχει τις αρχές αυτές για αυτού του είδους χρηστή διαχείριση. Έχει ένα ειδικό όργανο. Έχουμε και εμείς βέβαια τις απόψεις μας, αλλά δεν έχουμε δει και πάρα πολλές χώρες που θέλουν να τα εφαρμόσουν αυτά. με Μεταρρύθμιση που να εφαρμοστεί και να είναι υποχρεωτική. Ποιο θα πληρώνει αυτόν ο οποίο θα μελετάει το στοιχείο του κινδύνου, σε ποιον θα αναφέρεται το άτομο αυτό όσον αφορά όταν εντοπίζει κάποιο κίνδυνο κλπ. Για τη διαφάνεια έχουμε χώρε που λένε θα θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα όπου δεν έχουμε προϊόντα κεφαλαίου να τα χαρακτηρίσουμε διαφορετικά. Μα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χρηστή διαχείριση αν αρχίζετε να μεταμφιέζετε τα προϊόντα και να τους δίνετε διαφορετική παραπλανητική ονομασία. Αν είναι ένα προϊόν πιστοτικό θα πρέπει να έχει την ονομασία του, αν αναφέρεται στην αγορά πρέπει να έχει την ονομασία του, αν πάμε να την ανακατέψουμε δεν είναι πια χρηστή διαχείριση αυτή, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει πια Περί πρόκειται. Ξέρω ότι μιλάω τώρα, πετάγουμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά επειδή δεν έχω χρόνο θα σας πω. Αν έχουμε εταιρείε, ε, τράπεζες και θηγατρικές που ε, συνεργάζονται με επιχειρήσεις, αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό αύριο, να κάνουμε αυτό τον διαχωρισμό, και αυτό είναι μακρόπνος σχεδιασμός για την οικονομία, να φροντίσουμε τα κεφάλαια των ε, υποκαταστημάτων να είναι χωρισμένα, να ξέρει κάθε, η κάθε μονάδα τι κεφάλαιο διαθέτει, ούτως ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει σωστά. Ρωτήστε, τες, μιλήσετε, αναφερθήκατε στην εσωτερική αγορά. Αυτό σχετίζεται με αυτά που σας έλεγα τώρα δηλαδή για τη τοπική εποπτεία και να μην υπάρχει ένας επόπτης στο κέντρο, αλλά να υπάρχει εποπτεία και στις μικρές, στα υποκαταστήματα ή στις θεκατρικές. Επαναλαμβάνω λοιπόν, Μπορεί αυτά που λέμε να μην τα εισακούσει κανείς. Πάντως εμείς είμαστε υπέρ του να υπάρχει μια ευρύτερη εποπτική αρχή με βάση την δικαιοδοσία, μάλλον το νομικό καθεστώ στο οποίο λειτουργούν οι τράπεζες αυτές, επίσης να γίνεται και σε χαμηλότερο επίπεδο υποκαταστημάτων κλπ. ώστε να εξασφαλίζεται ότι υπάρχει παντού το αναγκαίο κεφάλαιο. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους. Ο κ. Σουάλτ από την Κομισιόν είναι παρόν. Δεν μπορώ να του δώσω το λόγο να απαντήσει όλα τα ερωτήματα, αλλά έχω ένα ερώτημα προς αυτόν τον ίδιο και νομίζω ότι όλοι μας θα θέλαμε να ακούσουμε, ιδίω οι σκιώδεις εισηγητές και ο εισηγητής για τα θέματα αυτά. Ακούσαμε από τον κύριο Βάλταο ότι η Επιτροπή της Βασιλείας περιμένει να συναρμοστούν όλα τα κομμάτια του παζλ τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο με την ε, αξιολόγηση αντικτύπου για να δουν πώς θα συγκεντρωθούν και θα συναρμοστούν όλα αυτά τα στοιχεία αυτά. Πώς θα τα λάβουμε εμείς αυτά υπόψη οι αλληλοεξαρτήσεις της ε, οδηγίας και τη φελογική επάρκεια 3 και 4. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να αντιμετωπίσουμε όλες τις πτυχές της 3. Ε, και όταν έχουμε τελειώσει όλα, όλη αυτή την αξιολόγηση βλέπουμε ότι η Επιτροπή της Βασιλείας έχει υποβάλει προτάσεις που εμείς δεν τις είχαμε φανταστεί. Τι θα κάνει η Κομισιόν για να τα αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πριν απαντήσω αυτό το ερώτημα, να σας δώσω και κάποια γενική εικόνα για το τι κάνουμε στην Επιτροπή. Μια επισκόπηση. Εμείς υποστηρίζουμε φυσικά την ατζέντα των G20 και το έργο της Επιτροπής Βασιλείας και εμείς συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με την Επιτροπή της Βασιλείας για όλα αυτά τα θέματα με στόχο να εξασφαλίσουμε ότι οποιασδήποτε ιδιαιτερότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποιασδήποτε διαφορές σε ό,τι αφορά τα επιχειρηματικά μοντέλα μας θα ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα τον αντίκτυπο και η Κομισιόν αποδίδει βέβαια τεράστια προσοχή στο θέμα της αξιολόγησης αντικτύπου για να μπορέσουμε να τονίσουμε, πόσο, να, να δείξει πόσο μεγάλη αυτή είναι η σημασία. Η Επιτροπή ζήτησε από την Επιτροπή Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις ε, εποπτών μάλλον, για τράπεζες να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους ε, επόπτες να καταλάβουν αν υπάρχουν ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες και ποιες είναι και οι επιπτώσεις αυτών των ιδιαιτερότητων. Και θέλω να τονίσω επίση και τη σημασία της διαδικασίας διαβούλευσης. Θέλουμε να κατανοήσουμε ποιες είναι αυτές οι ιδιαιτερότητες. Γι' αυτό η Κομισιό ξεκίνησε μια διαδικασία διαβούλευσης παράλληλα με την διαδικασία της Λειτουργίας Επιτροπής της Βασιλείας. Οργανώσαμε και μια δημόσια ακρόαση, η οποία έλαβε χώρα την προηγούμενη Δευτέρα, την προηγούμενη εβδομάδα και είχαμε πάνω από 150 συμμετέχοντες, ουσιαστικά όλους τους σημαντικούς εμπλεκόμενους στον τομέα αυτό που θέλαν να λάβουν το λόγο είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, εμείς προβλέπουμε να έχουμε κάποια προκατακτικά αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης αντικτύπου το καλοκαίρι, οπότε πράγματι είναι κάτι το οποίο ευθυγραμμίζεται με τη διαδικασία της Βασιλείας και η Κομισιόν επίσης αποδίδει μεγάλη σημασία στο να υπάρξει μια ανάλυση μακροοικονομικού αντικτύπου και γι' αυτό κάνουμε αυτή την εσωτερική ανάλυση με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και εμπειρογνωμόνων από άλλες γενικές διευθύνσεις που θα αντιμετωπίσουν αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα. Κλείνοντας, θέλω να κάνω μια σημαντική ε, παρατήρηση που έχει να κάνει με τη διαφάνεια και την θέληση συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πολλέ από αυτέ τι προτάσει μπορεί να έχουν ένα πάρα πολύ σοβαρό αντίκτυπο. Ένα από τα στοιχεία που δείχνει αυτή τη θέληση συνεργασίας είναι η διαβούλευση που ξεκινήσαμε τον Φεβρουάριο και η δημόσια ακρόαση που οργανώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαστε έτοιμοι και ανοιχτοί να ακούσουμε όλες τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων. Δεν έχει ακόμα ληφθεί κάποια απόφαση προς το παρόν. Θα πρέπει να καταλάβουμε αν υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής ε, πλευράς που πρέπει να αντανακλώνται στην τελική πρόταση και αυτά θα ήθελα εγώ να πω από τη δική μου πλευρά από την Κομισιόν. Αν έχετε κάποια ερωτήματα που θέλω να απαντήσω, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Όχι, όχι, λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι ήδη έχω ξεπεράσει την ε, γενεοδορία των εισηγητών για τα επόμενα θέματα στην μέση διάταξη. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ. Νομίζω ότι πολλοί από εμά ακόμα είμαστε σε αβεβαιότητα για το πώς θα πρέπει να περατωθεί αυτή η διαδικασία και πώς θα πρέπει να περατώσουμε μια νομοθετική πρόταση και την αξιολόγησή της όταν δεν έχουμε ακόμα τις μελέτες αντικτύπου. Η εξέταση της, του σχεδίου έκθεσης του κ. Κάρας θα γίνει την 1η Ιουνίου Στη συνέχεια προβλέπουμε να έχουμε μια πρόθεση για τροπολογίες 8 Ιουνίου, να εξεταστούν μετά στις 28 Ιουνίου όταν ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε στις 6 Σεπτεμβρίου ως Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων. αυτό είναι το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την έκθεση του κυρίου Καράς για τη κεφαλουργική επάρχεια 4. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ όλους τους ομιλητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν και βλέπω ότι υπήρξε και επαφή με τους βουλευτές ανταλλάσσετε επισκεπτήρια ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση και στο μέλλον. Τώρα, δύο λεπτά διάλειμμα για να φύγουν αυτοί που θέλουν να φύγουν. Παρακαλώ, όσοι θέλετε να φύγετε, να το κάνετε με ηρεμία και ησυχία, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα και να δώσουμε τη δυνατότητα στον Hans Peter Μάρτιν να έχει κάποιο γαλήνιο περιβάλλον να παρουσιάσει την πρότασή του. Όσοι δεν θέλουν λοιπόν να μείνουν, παρακαλώ να φύγουν με ταχύτητα και γαλήνη. Um, could παρακαλώ πολύ γιατί έχουμε δύο ακόμα σημεία στη μερίσια διάταξη. Περνάμε στο σημείο 4. Σας παρακαλώ πολύ αν θέλετε να συζητήσετε με κάποιον κάντε το εκτός εθούσης. Πρέπει τώρα να δώσω το λόγο στον Hans Peter Martin για να μας μιλήσει για το σχέδιο γνωμοδότησής του για την διασύνδεση των μητρών επιχειρήσεων. Κύριε Μάρτιν, μπορείτε να μιλήσετε τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να είμαι πολύ σύντομο. Και ενώ είναι πάρα πολύ αφηρημένα αυτά τα θέματα και σας φαίνονται υπερβολικά τεχνικά και αφηρημένα, έχουν μεγάλη σχέση με θέματα που μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το έλλειμμα πληροφορία σε ό,τι αφορά τις χρηματαγορές και τις επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις. Η πράσινη βίβλωση Κομισιόν αναφέρεται στο θέμα αυτό τα μητρώα επιχειρήσεων πρέπει να συνδέονται καλύτερα στο μέλλον και να υπάρχει το νομικό πλαίσιο να αντιμετωπίσει κείμενη διαδικτύωση αυτών των μητρώων που λειτουργούν πια ηλεκτρονικά σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε διαμεθοριακό επίπεδο. Ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε να υπάρξει η απαραίτητη ανάπτυξη και στην εσωτερική αγορά επί τη βάση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ώστε να αντιμετωπίσετε η περίπτωση επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν σε ένα κράτος μέλος αλλά είναι δραστηριοποιημένες και σε άλλα κράτη-μέλη. Όλα αυτά είναι σημαντικά και για τον ε, καταναλωτή αλλά και γενικά για την ασφάλεια δικαίου. Η λεγόμενη ομάδα Stoiber έχει ξεκινήσει ήδη να εξετάζει το θέμα αυτό και θεωρούν ότι με μια πιο αποτελεσματική ε, διασύνδεση των ευρωπαϊκών μητρών επιχειρήσεων θα μπορέσουμε να έχουμε μια σημαντική εξοικονόμηση που θα είναι εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ. Εγώ δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με αυτά τα οποία έχουμε ενώπιόν μας. Υπάρχει η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μητρών, αλλά συγχρόνως υπάρχει και ένας εθελοντικός χαρακτήρας ο οποίος συναρμόζεται με μια πάρα πολύ πολύπλοκη διαδικασία. Ένα άλλο, μια άλλη πρόταση είναι το να υπάρξει η διαλειτουργικότητα των μητρών και αυτό είναι μια ερευνητική, μια ερευνητική ε, ενέργεια που δεν έχουμε ακόμα αποτιμήσει τα αποτελέσματα. Και υπάρχει και το σύστημα IMI το οποίο αφορά περισσότερο την παροχή υπηρεσιών μέσα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για την δικαιοσύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχει να κάνει με την ανταλλαγή πληροφοριών σε δικαστικές διαδικασίες. Το ερώτημα πάντως που μας απασχολεί είναι κυρίως πώς οι πληροφορίες είναι η πληροφορίες για ιδρύματα εγγεγραμμένα στα χρηματιστήρια μπορούν να είναι εύκολα προσβάσιμες στους πολίτες, τους καταναλωτές και τους επενδύσεις. Και φυσικά θα πρέπει να ληφθεί μέσα στο πλαίσιο αυτό η ανάγκη να υπάρξει αποδοτικότητα και διαφάνεια όπως έχει τονίσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η Κομισιόν μας ρωτάει αν θέλουμε περισσότερα μητρώα επιχειρήσεων Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι ναι για να έχουμε και μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Θέλουμε ένα σύστημα ολοκληρωμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο θα μειώσει τη γραφειοκρατία αλλά δεν θέλουμε να εκθέσουμε ε, σε κινδύνους το σύστημα προστασίας των δεδομένων, των ευαίσθητων δεδομένων των επιχειρήσεων. Αυτά ήθελα να πω λοιπόν και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και εάν κάποιος θέλει να παρέμβει είμαι έτοιμος να απαντήσω και να ακούσω τις ε, απόψεις και τις εκτιμήσεις των συναδέλφων για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντικαθιστώ εδώ το δικό μας σκιώδη ηγητή τον κύριο Πίτερ Ζήμων, ο οποίο ασχολείται με το θέμα αυτό, η άποψή μα, είναι ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο μέσα στο νομοθετικό πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα σημαντικό κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Το ότι δεν υπάρχει μια δυνατότητα να έχει κανεί ένα ενιαίο μητρό επιχειρήσεων. Αυτό είναι σημαντικό και για τις επιχειρήσεις και για τους πιστοτικούς φορείς, αλλά ουσιαστικά είναι σημαντικό και για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Θα σας υπενθυμίσω πόσο μεγάλες είναι οι δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν στην πρακτική εφαρμογή της <clears throat> οδηγίας για την παροχή υπηρεσιών όταν δεν ξέρουμε ποια είναι η εταιρεία με την οποία έχουμε να κάνουμε ως πάροχο υπηρεσιών, κατά πόσο λοιπόν μπορούμε να έχουμε αυτές τις πληροφορίες με αξιόπιστο τρόπο και χωρίς υπερβολική γραφειοκρατία για να ξέρουν οι επιχειρήσεις με ποιους συναλλάσσονται, αυτό θα ήταν πάρα πολύ θετικό. Υποστηρίζω λοιπόν αυτά που λέει ο συγητής. Ναι, πράγματι θέλουμε να υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο να έχει και υποχρεωτικό χαρακτήρα και εδώ υποστηρίζουμε την Κομισιόν. Μόνο έτσι έχει νόημα, δεν μπορεί να είναι εθελοντικού χαρακτήρα, πρέπει να είναι υποχρεωτική η παρουσία σε αυτό το σύστημα, πρέπει να είναι επίσης αποτελεσματικό. Δεν θέλουμε εμείς να αυξήσουμε την ε, γραφειοκρατικότητα. Θα πρέπει όμως να υπάρχει δυνατότητα να ελέγχει κανείς το περιεχόμενο του, θα πρέπει να είναι αναγνώσιμο και επομένως θα πρέπει να, να περιλαμβάνει και σωστή προστασία των ε, δεδομένων. Μέσα στα πλαίσια αυτά εμείς ε, υποστηρίζουμε αυτή την πρόταση η οποία τονίζω και πάλι θα κλείσει ένα σημαντικό κενό στην εσωτερική αγορά. Κάποιος άλλος θα ήθελε να λάβει το λόγο. Κύριο Σουάμπ. Ευχαριστώ και εγώ κυρία Πρόεδρε. Ίσως μπορώ να προσθέσω κάτι το οποίο ήταν σημαντικό για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ότι υπάρχει η ανάγκη να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία αυτού του Μητρώου Επιχειρήσεων. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα υπήρξε κάποιο πρόβλημα με το θέμα της εισαγωγής των επιχειρήσεων στα θέματα αυτά, αλλά νομίζω θα ξε... η πρωτοβουλία αυτής της Κομισιόν θα αυξήσει σημαντικά την αξιοπιστία αυτού, του, αυτών των μητρών και κυρίως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια σε διαμεθοριακό επίπεδο και γι' αυτό εμείς υποστηρίζουμε εν, ένθερμα αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ, λέει κύριε Πρόεδρος. Εγώ είμαι σκιώδης συζητήτρια για τη δική μου ομάδα και από κάποιες απόψεις θεωρώ ότι αυτή η πρόταση συνδέεται με αυτά τα οποία κάναμε στην προηγούμενη θητεία όταν αναφερόμαστε για το καταστατικό για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία όταν το <clears throat> εκπονούσαμε αυτό το, το, το νομοθέτημα, μας ενδιαφέρει τι γίνεται με επιχειρήσεις που έχουν την κεντρική τους έδρα σε μία χώρα, αλλά το γραφείο τους εκεί που είναι καταγεγραμμένη επιχείρηση βρίσκεται σε άλλη χώρα. Θέλαμε να εξασφαλίσουμε λοιπόν να υπάρξει μια διασύνδεση των πληροφοριών, ώστε να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση και από τις δύο αυτές τοποθεσίες και μας ενδιέφερε ιδίως η ιδέα του να υπάρχει ένα κεντρικό ευρωπαϊκό μητρό, να υπάρχει δυνατότητα να κατατίθενται ε, έγγραφα σε αυτό το κεντρικό επίπεδο. Δεν θέλαμε να, θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι η υποβολή εγγράφων στο κεντρικό μητρό δεν θα, έκανε, ε, θα αφαιρούσε την ανάγκη να υπάρχει και υποβολή τους στα τοπικά γραφεία των επιχειρήσεων. Δηλαδή θα μειώναμε την ε, γραφειοκρατία. Το βασικό είναι να υπάρχει ένας βασικός τόπος όπου μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα μιας επιχείρησης. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απαραίτητο φυσικά όλα αυτά τα στοιχεία να είναι προσβάσιμα σε δημόσιο επίπεδο. Και σε ό,τι αφορά το εφικτό ή όχι ενό τέτοιου συστήματο. Φυσικά θα υπήρχαν ορισμένε πτυχέ προστασία δεδομένων οι οποίε θα εφαρμοζόντουσαν. Συνήθω μιλάμε για έγγραφα τα οποία είναι διαθέσιμα σε ένα κράτο μέλο και δεν καταλαβαίνουμε ότι κάτι που είναι διαθέσιμο σε ένα κράτο μέλο δεν μπορεί να είναι διαθέσιμο με τον ίδιο τρόπο και σε άλλα κράτη-μέλη. Γιατί λοιπόν πρέπει να εφαρμόζεται η προστασία δεδομένων που να αφορά του πολίτε άλλων κρατών μελών. Θα πρέπει και αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να τα εξετάσουν και να αναδυφίσουν αυτά τα έγγραφα. Δεν θέλω βέβαια να μπούμε τώρα σε προβλήματα θεωρώντας ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο. Βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια ενιαία αγορά. Κάτι το οποίο είναι προσβάσιμο βάσει των κανόνων μιας χώρας μέλους θα πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτά ήθελα να πω λοιπόν προς το παρόν και θα επανέλθω στο θέμα αυτό όταν πρέπει να καταθέσουμε τροπολογίες και που φανταζούμε θα εκπνεύσει σύντομα η προθεσμία της τροπολογίας. Κύριε Μάρτιν, θέλετε να πείτε κάτι. βεβαίω. Θέλω να ευχαριστήσω, για τις... Ε, Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για, την, ε, για τις προτάσεις τους. Θέλω να τονίσω λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Μπούλμαν, ότι πρέπει να είναι κάτι το οποίο είναι αποτελεσματικό, διάφανο, υποχρεωτικό και μειώνει τη γραφειοκρατία και ίσως μπορεί και η γραμματεία να με βοηθήσει να τα διατυπώσω όλα αυτά με καλύτερο τρόπο, αυτά τα οποία σας λέω λιγάκι τηλεγραφικά. Για αυτά που είπατε κύριε Σφαμπ, θα ήταν πολύ όμορφο, να, όπως είπε και η πρόεδρος, αν όλα τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα σε μια χώρα να είναι διαθέσιμα σε όλες τις άλλες χώρες υπήρξε μια περίπτωση που ήταν κάποια στοιχεία τα οποία έδωσε το Συμβούλιο και η Κομισιόν για μια επιχείρηση τα οποία μπορούσαν να τα έχουν όλοι, αλλά κυρία Μπόουλς υπήρχαν πολλά τέτοια έγγραφα τα οποία δεν μπορούμε να τα παίρνουμε με την ευκολία που θα θέλαμε να έχουμε, αλλά σίγουρα να γίνει κάτι τέτοιο αυτό θα οδηγούσε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για τις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η προθεσμία είναι η 10η Μαΐου το μεσημέρι, στο 12 το μεσημέρι για την υποβολή τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε στις 2 Ιουνίου αφού συζητήσουμε την πρώτη Ιουνίου της τροπολογίας και στις 23 Ιουνίου θα γίνει ψηφοφορία στην α, επί της ουσίας Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Υποβολή τροπολογιών λοιπόν μέχρι τις 10 Μαΐου σας παρακαλώ. Ας περάσουμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, υπαριθμών 5. Σχέδιο προπολογισμού 2011, όλα τα τμήματα και συντάξει γνωμοδότηση του Αντρέα Σουάμπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Το προηγούμενο σημείο διεκπαιρεώθηκε πολύ γρήγορα και θα προσπαθήσω και αυτό να κάνω το ίδιο. Θα ήθελα να σας πω καταρχήν ότι υπάρχει μια νέα διαδικασία η οποία εφαρμόζεται με την συνθήκη της Λισαβόνας. Επομένως, η διαδικασία του προϋπολογισμού είναι μια ειδική διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο σε μία ανάγνωση αποφασίζουν για τον ετήσιο προϋπολογισμό. Είναι η πρώτη φορά, η πρώτη χρονιά που εφαρμόζεται αυτή η νέα στρατηγική μετά την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας και δεν ξέρουμε αν αυτό θα αποδειχθεί επωφελές ή όχι, αλλά σίγουρα και εγώ και η Γραμματεία προσπαθήσουμε να μπορέσουμε να αποκομίσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα ενώπιον αυτής της πρόκλησης. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι αυτή η οποία είναι αρμόδια για αυτή την πρόταση. Στις 10 Μαΐου θα παρουσιάσει η συγγήτρια μια έκθεση για το τμήμα 3 του προϋπολογισμού. Οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 12 Μαΐου. Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα λοιπόν που έχουμε στη διάθεσή μας. Λόγω της επιταχυμένης αυτής της διαδικασίας και ίσως η γραμματεία τα ξέρει καλύτερα, και λέει εδώ το έγγραφό μου πρέπει οι τροπολογίε να πάνε κατευθείαν στην εισηγήτρια. Ελπίζω ότι αυτό. Στον εισηγητή δεν πιστεύω ότι αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερο φόρτο εργασία για μένα. Κάποια σημεία περιεχομένου. Τα ζητήματα όπου η Επιτροπή Οικονομικών και ε, Νομισματικών Θεμάτων θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά. Είναι θέματα που έχουν να κάνουν με τη στατιστική, το ζήτημα του, της Ευρωομάδος, η εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης όταν πρόκειται για θέματα προσωπικού, για φορολογία, η Κομισιόν έχει εμποδιστεί από το Συμβούλιο στο να καταρτήσει ένα πλήρη κατάλογο και αυτά θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά από το 2011. Είναι θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια και τη σταθερότητα στις χρηματαγορές. Η άλλη θέση είναι η προώθηση ευνοϊκότερη θέση για τις μικροπιστώσει στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι κανείς από μας γνωρίζει όλο τον προϋπολογισμό και έχει διαβάσει όλα αυτά τα θέματα, ε, δεν πρόκειται να σας ε, κουράσω με τις λεπτομέρειες, απλώς ε, έχουν καθοριστεί τα κονδύλια για την 7 περίοδο και απλώς θα υπάρξουν μικρές αναδιαθρώσεις και αναδιατυπώσεις από χρόνο σε χρόνο και πιστεύω ότι αν συμφωνείτε μαζί μου θα πρέπει να προσπαθήσουμε οι γραμμές του προϋπολογισμού να παραμείνουν στο επίπεδο του περσινού έτους και εάν χρειαστεί να κάνουμε κάποια τροποποίηση στο μέλλον, να εστιάσουμε την προσοχή μας στις, προετοιμασί... στις προτεραιότητες και φυσικά θα παραμείνω σε επαφή με τους σκιώδεις εισηγητές για τη δική μου άποψη. Εγώ νομίζω πρέπει να ενισχύσουμε ιδιαίτερα το έργο μας για τις στατιστικές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Thank uh, Σας ευχαριστούμε πολύ, Λουτβίξον. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέπουμε εδώ ότι η νέα διαδικασία πρόκειται να αλλάξει τη δυναμική της όλης διαδικασίας. Αν θέλουμε πραγματικά να πειράσουμε το τελικό αποτέλεσμα, τότε θα πρέπει να λάβουμε δράση πολύ νωρί στη διαδικασία. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό μέσω της Επιτροπής Οικονομικών, Οικονομικής και Μεσματικής Πολιτικής να καθορίσουμε ποια είναι η θέση μας και να λάβουμε δράση πολύ νωρίς. Πρέπει να μιλήσουμε με μία ενιαία φωνή στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πειράσουμε τα πράγματα καλύτερα αν είμαστε ενωμένοι από την αρχή. Σε μια αρχική φάση λοιπόν θα πρέπει να καταφέρουμε να πετύχουμε πολιτική συνένεση ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές ομάδες προκειμένου να δώσουμε μια κοινή απάντηση εξ ονόματος της Επιτροπής μας όσον αφορά το, σχέδιο, το προσχέδιο προπολογισμού του 2011 που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από μια πρώτη πολύ θετική συνάντηση που είχαμε με το στάκτη νομοδοτηση, θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτή την ε, πολύτιμη πολιτική συνένεση. Όσον αφορά τώρα τις γενικότερες εντυπώσεις από τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλύπτονται τα περισσότερα πράγματα πιστεύω. Υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία θα πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις, αλλά θα έλεγα σε γενικές γραμμές ότι το μεγαλύτερο τμήμα των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να γίνει αποδεκτό. Όσον αφορά τώρα το σύνολο του σχεδίου προπολογισμού, πιστεύω ότι υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, το περιθώριο στο κεφάλαιο 1α είναι πολύ στενό, μολονότι εδώ πέρα υπάρχει μια αύξηση στο σχέδιο προπολογισμού όσον αφορά το αρχικό σχέδιο. 50,1 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό το οποίο προβλέπεται αυτή τη στιγμή και το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ χαμηλό. Το πολύ μικρό αυτό περιορισμένο περιθώριο δεν πρόκειται να μας δώσει κανένα, καμία δυνατότητα ελιγμού για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση και να εφαρμόσουμε το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης. Μολονότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντιδράσει αρνητικά, πιστεύω ότι θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση προκειμένου να αυξηθεί η συγκεκριμένη γραμμή του προπολογισμού. Ένα δεύτερο τώρα σημείο. Η άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής του 2020. Έχω κάποιε αμφιβολίε για την στάση που κρατά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθότι δεν μα έχει δώσει κανένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για την χρηματοδότηση αυτή στρατηγική. Ουσιαστικά χρησιμοποιεί τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα και αυτό για μένα είναι πρόβλημα. Είμαι πεπισμένος ότι ε, χρειαζόμαστε νέα κονδύλια για τις νέες αυτές πρωτοβουλίες. Αυτό είναι εκ των, των ουκάνευ, προκειμένου να καταφέρουμε να βάλουμε σωστό δρόμο τη νέα στρατηγική. Επίσης, η στρατηγική αυτή του 2020 χρηματοδοτείται κυρίως υπό την ε, κατηγορία 1α, το κεφάλαιο 1α και στο σημείο αυτό συνδέεται η στρατηγική αυτή με το πρόβλημα το οποίο ανέφερα πριν από λίγο. Ούτε για τη στρατηγική αυτή υπάρχει κάποιο περιθώριο αύξηση των κονδυλίων και επομένω δεν υπάρχει περιθώριο ελιγμών. Πρέπει να στείλουμε ένα σαφέ μήνυμα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προ το Συμβούλιο. Αν δεν έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια για να εφαρμόσουμε τη στρατηγική του 2020, τότε ίσω να, μην είναι αξιόπιστη στο τέλο αυτή η στρατηγική. και βέβαια οι καλές προθέσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από συγκεκριμένε πράξεις και ουσιαστικά χρηματοδότηση. Επίσης βλέπουμε κάποια μείωση των χρηματοδοτικών μέσων που έχει να κάνει με το συντονισμό της εσωτερικής αγοράς. Βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικές διακοιμάνσεις αυτή τη στιγμή στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Πιστεύω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να δυναμώσουμε τις δραστηριότητές μας και όχι να τις μειώσουμε. Υπάρχει εδώ μια γενικότερη ε, αύξηση. Παρόλα αυτά δεν μπορώ να υποστηρίξω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε μειώσει σε κάποια σημεία, τις οποίες θα πρέπει να συζητήσουμε. Πρέπει να δούμε αν είναι δυνατόν να ενδυναμώσουμε τα όσα προβλέπονται στον προπολογισμό για, τα, για τις στατιστικές. Τα τελευταία γεγονότα καταδεικνύουν ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς πρόσβαση σε αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά και τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Όσον αφορά τα τελωνία και τα φορολογικά ζητήματα, δεν μπορώ να υποστηρίξω πάλι το σχέδιο προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθότι δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη αύξηση των κονδυλίων για την διεθνή συνεργασία. Μια θετική πτυχή βέβαια στο σχέδιο προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι ε, γίνεται μία πρόταση στο κεφάλαιο 2 για 50 εκατομμύρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το υφιστάμενο εδώ περιθώριο προκειμένου να καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε την ε, νέα αυτή υπηρεσία εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα θετικό ακόμα στοιχείο είναι η αύξηση προτείνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολιτική ανταγωνισμού. Σε οικονομικά δύσκολε εποχές χρειαζόμαστε στεναρά μέτρα εξ ονόματο Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, περισσότερο σήμερα από ό,τι ποτέ. Συνοψίζοντα, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε. Το σχέδιο προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν περιέχει κάποιε εκπλήξει ούτε μεγάλε ανισορροπίε τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, από την εξ τη της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής. Ο κύριος Κάρας έχει το λόγο. Κύριε Σιγητά, θα ήθελα και εγώ να τονίσω ότι η Κομισιόν με τις νέες ρυθμίσεις δεν έχει κανένα περιθώριο ελιγμών για σημαντικά θέματα. Πρέπει να δημιουργήσουμε και κάποιο περιθώριο ελιγμών για την Κομισιόν για να μπορούμε να ασχολούμαστε με πολιτικές λύσεις και να μην είμαστε απλώς μια μηχανή διανομής τράπουλας. Επίσης, οι στόχοι της Ευρώπης 2020, Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα εργαλεία του προπολογισμού. Γι' αυτό ο προπολογισμό του 2011 ήδη θα πρέπει να αντανακλά την στρατηγική τη Ευρώπη 2020 και δεν μπορεί να είναι απλώ status quo. Τρίτον, έχουμε δύο σημαντικά στοιχεία στην στρατηγική της Ευρώπης 2020 που να αποτελούν και απάντηση στην κρίση που αντιμετωπίζουμε. Χρειαζόμαστε περισσότερα ευρωπαϊκά σχέδια σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, την καινοτομία, την έρευνα και την κατάρτιση για να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν τα πράγματα αν εμείς έχουμε απλώς τους, υπο, τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών σε μια αθρηστική διαδικασία θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ένα πρωτοπόρο ρόλο για την, για την χρήση των πόρων σε αυτή την κατεύθυνση. Το επόμενο σημείο αφορά την Eurostat και αυτά που είπατε προηγουμένως αν στην περίπτωση κρίσεων όπως αυτής που έχουμε με την ε, Ελλάδα τώρα, αν θέλουμε να έχουμε καλύτερο έλεγχο για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εφαρμογή των κανόνων, χρειαζόμαστε να έχουμε ένα ανεξάρτητο χρηματο, ε, στατιστικό φορέα, τη Eurostat, ο οποίο θα έχει του απαραίτητου οικονομικού πόρου και το απαραίτητο προσωπικό. Και αυτό θα πρέπει να καταγραφεί και στον προπολογισμό του 2011 γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε την πολιτική μας αξιοπιστία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των πολιτικών μας προτεραιοτήτων. Ευχαριστώ. Κύριε Κλούτ. Σας ευχαριστώ. Και εμένα μου άρεσε βλέποντας τα αριθμητικά στοιχεία ότι υπάρχει μία περισσότερο από αναλογική αύξηση του προπολογισμού στον τομέα τη εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Αλλά αυτό θέτει το θεμελιώδες πρόβλημα από τη δική τη πολιτική ομάδα, βέβαια, αν αυτό είναι απαραίτητο και αν αυτό βοηθάει να δημιουργήσουμε και τις υποδομές ε, που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη απασχόληση και την αντιμετώπιση της ε, ένδυα και του κοινωνικού αποκλεισμού που βλέπουμε. Αν μπορούν όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν να πραγματοποιηθούν. Αν θέλουμε να το κάνουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να κάνουμε και περισσότερα πράγματα από αυτά που έχουμε κάνει εφέτο. Θα πρέπει να υπάρξουν επενδύσει προ την κατεύθυνση αυτή, όπω είπε και ο προλαλή σα. Θα ήθελα να εξασφαλίσω ότι δεν θα πάνε όλα αυτά τα χρήματα στην εξωτερική πολιτική, γιατί βλέπω εκεί πέρα μια υπέρμετρη και όχι αναλογική αύξηση του προπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρο. Δεν θέλει κανεί να λάβει το λόγο. Ο κύριο Σουάπ και πάλι. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Σουάπ. Πάρα πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ καταρχήν τους συναδέλφους για τις ε, ε, προτάσεις τους και τη συμβολή τους στη συζήτηση. Θα ήθελα να απαντήσω στον Σουηδό μου συνάδελφο από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Θέλω να υπάρχει μια κοινή πρόταση για τον προϋπολογισμό η οποία να ξεπερνάει τις παραταξιακές θέσεις και είμαι έτοιμος να συνεργαστώ μαζί σας και είμαι ευγνώμων για τις προτάσεις σας, για τα... τις προτάσεις του Ότμαρ Κάρας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Θα πρέπει η Κομισιόν να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τις πολιτικές τις οποίες έχουμε θεσπίσει και γι' αυτό η στατική της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης για το 2020 θα πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί για τον κύριο Κλούτερ και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε ότι αυτή τη στιγμή είναι υψηλότερος ο προϋπολογισμός για τα θέματα ασφάλειας και εξωτερικής, ε, εξωτερικής πολιτικής, αλλά βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη για τα θέματα αυτά. Σε άλλες θέσεις του προϋπολογισμού εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι υπάρχουν πολλοί τομεί οι οποίοι δεν είναι επαρκού χρηματοδότηση για θέματα τα οποία για μα είναι προτεραιότητες και θα το τονίσω αυτό και ενώπιον του Συμβουλίου. Αυτά είναι από τη δική μου πλευρά. Κυρία Πρόεδρε, εγώ θα συνεργαστώ με του ε, σκιώδεις εισηγητές από τι άλλε πολιτικέ ομάδε για να μπορώ να σα φέρω το ταχύτερο δυνατόν μια πρόταση και μετά εναπόκειται σε εσά και την γραμματεία και τους συντονιστές να μπορέσουμε να δούμε πώς θα γίνει η συνέχεια των εργασιών μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει και Πρόεδρος. Λοιπόν, έχουμε την ε, εξέταση του σχεδίου γνωμοδότης 21 Ιουνίου, 19 Ιουλίου προθεσμία για τροπολογίες, η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 6 Σεπτεμβρίου και η κύρια Επιτροπή στις 20 Σεπτεμβρίου και θα πάμε μάλλον στην ε, δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου. Αυτά είναι η πρόβλεψη προς το παρόν σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα αυτής της έκθεσης και όλα αυτά φέρνουν την απογευματινή μας συνεδρίαση σε ένα πέρας. Όπως είπα και στην αρχή, δεν έχουμε την παρουσία της κυρίας Σαλγκάδου αύριο το πρωί, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε το χρόνο από τις 9.30 και μετά για να κάνουμε μια συζήτηση μεταξύ μας στην Επιτροπή αυτή για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της Ελλάδος και άλλα ζητήματα τα οποία μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και φυσικά στη συνέχεια θα είναι παρόν και ο Επίτροπος ε, Μπάρνιε. Νομίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή προθέρμανση πριν συναντήσουμε τον κύριο Μπαρνιέ. Σας ευχαριστώ όλους και θα τα πούμε αύριο το πρωί.